Uh, um, uh, Καλημέρα σας όλοι. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους ε, τη λιμένη αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που είναι τόσοι πολλοί παρόντες. Uh, Ελπίζω κάποιοι από συναδέλφους μου να έρθουν σε λίγο. Αλλά είναι ώρα νομίζω να αρχίσουμε. Γιατί έχουμε την τύχη να έχουμε την Επίτροπο Vivian για δικαιοσύνη, βασικά δικαιώματα και τον Τζονταλή μαζί μας που είναι για τα θέματα της δημόσιας υγείας. <clears throat> Σε αυτή την κοινή ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία ακρόαση για το πάρα πολύ σημαντικό θέμα της ατζέντα για τον καταναλωτή 2014-2020. Η Επίτροπη Ρέντιν και Ντάλι εργάζονται από κοινού πάνω σε αυτό και προβλέπουμε βέβαια να δούμε το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Θα μας δώσουν ίσως κάποιες ενδείξεις πότε θα ετοιμαστεί η πρόταση. Ίσως κάποιες ιδέες που θα δοθούν σήμερα θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έντονα υποστήριξε δική μας ε, ε, Επιτροπή και, και χαιρετίζω τον κυρία Τρενταφυλλίδη που ήταν εισηγητής της δικής μας έκθεσης ε, για το τι πιστεύουμε θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η ατζέντα και θα του δώσω το λόγο μετά που θα κάνουμε τον πρώτο γύρο συζητήσεων με τους Επίτροπους. Η Επιτροπή είναι μαζί μας μέχρι τις 10 και θα δεχθούν και ερωτήσεις και χαιρετίζω επίσης τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Δανίας, τον κύριο Νίσπορκ, που ασχολήθηκε πάρα πολύ με την εργασία μας. Σας χαιρετίζουμε λοιπόν. Είναι καλό λοιπόν που έχουμε και εκπροσώπηση του Συμβουλίου εδώ και θα του δώσω επίσης το λόγο και πράγματι η Δανική Προεδρία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την προώθηση της ε, πολιτικής για τους καταναλωτές και θα οργανώσει μια παγκόσμια ημερίδα για τους καταναλωτές προσεχώς. Θα δώσω το λόγο καταρχήν τους επιτρόπους στον ε, μόνιμο αντιπρόσωπο και μετά θα σας ε, ε, δώσω δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήσεις. Θα δεχτώ ερωτήσει από όλους. Αν θέλει λοιπόν κάποιος να υπο... στείλει ένα σημείωμα, ότι θέλει να πάρει το λόγο να υποβάλει μια ερώτηση, να το στείλετε. Και θέλω να σας υπενθυμίσω όλους ε, ότι το, η συνεδρία σε αυτή περνάει στο διαδίκτυο και να χαιρετήσω και όλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή στο web stream. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ καλό για μας να υπάρχει αυτή η διαφάνεια. Καλωσορίζω λοιπόν όλους τους ακροατές. Uh, και εάν έχετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, στείλετε ένα email στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οπωσδήποτε θα ληφθεί υπόψη. Θα δώσω τώρα αμέσω ε, στη Vivian Redding. Σα χαιρετίζουμε. Είσαστε συχνά στο Κοινοβούλιο. Σα χαιρετίζουμε σε αυτή τη συνεδρίαση και θα σα δώσω το λόγο για να μα κάνετε μια πρώτη παρουσίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα χαιρετίζω, κυρίε και κύριοι. Ο συνάδελφο Τζονταλή και εγώ ε, ασχολούμεθα από κοινού πάνω στο θέμα αυτή της ατζέντα κατανοητή, αλλά ο Τζον θα σας παρουσιάσει τις λεπτομέρειες το τι προετοιμάζουμε. Θα σας πω δύο λόγια του το τι έχουμε κατά νου αυτή τη στιγμή που είναι η οικονομική κρίση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στην κρίση αυτή να δράσουμε για να ενθαρρύνουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά. Γιατί μόνο ε, που έχουν εμπιστοσύνη μπορούν να ενθαρρύνουν τη ζήτηση που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη που χρειαζόμαστε. Έχουμε τεράστιο δυναμικό στην ενιαία αγορά. Δυναμικό όμως που δεν τη χάνει πλήρης εκμετάλλευση, όπως θα έπρεπε. Παράδειγμα, ε, οι αγορές online ε, διαμεθοριακά παρουσιάζουν 16% 16 φορές περισσότερα προϊόντα για επιλογή, αλλά 60%, 60 των ίσων των καταναλωτών δεν χρησιμοποιούν την δυνατότητα αυτή και γιατί, γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη του τι γίνεται όταν ψωνίζουν έτσι με το διαδίκτυο σε μια άλλη χώρα. Λοιπόν, η δημιουργία της εμπιστοσύνη είναι η πρώτη μας ε, προτεραιότητα. Και έχοντας κατά νου τις προτεραιότητες, έχω και κατά νου τον κόσμο των ψηφιακών προϊόντων που εμπλουτίζει τη ζωή μας, που συμβάλλει στην, στην οικονομία των χωρών μας. Παρ' αυτά και εδώ υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Ποιος από σας ε, δεν ε, ε, έκρισε ένα κουτάκι στο διαδίκιο χωρίς να ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειτο και τι α, ευθύνες ανέλαμβανε ή ποιο από εσά ξέρει ακριβώς σε ποιον θα πρέπει να παραπονηθεί εάν κάτι δεν πάει καλά με την, μια αγορά στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα αυτών των ε, δεδομένων είναι πολύ γνωστά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο ιστορικό της Ένωσης είναι λιγότερο από 5% των ε, πωλήσεων λιανικής ε, αγοράς. Και πάνω από το 50% των καταναλωτών έχουν κάποια προβλήματα πάντα όταν χρησιμοποιούν αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε καλύτερη προστασία για τα παιδιά μας επίσης και άλλους ευάλωτους καταναλωτές στο διαδίκτυο. Ξέρετε ότι υπάρχει ε, το κεκτημένο για την ε, προστασία των καταναλωτών, υπάρχουν σχετικοί κανόνες όποτε είναι ε, θύματα θέμη των ε, πρακτικών ή όταν αγοράζουν κάτι. Πέρσι έχουμε την ε, οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και όταν μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια θα ενδυναμώσει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ορίζοντας παραδείγματος χάρη ομοιόμορφα χρονικά όρια για τα, για τα συμβόλαια αυτή ή όσον αφορά το κόστος των πωλήσεων οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τον νομικό κατακαιρματισμό των ε, αγορών, δίνοντας τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ένα ενιαίο νόμο πωλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ένα πρόσφατο σχέδιο τη δέσμη για την αναθεώρηση της προστασίας των δεδομένων, που θα ενδυναμώσει τα σχετικά δικαιώματα των καταναλωτών, ιδίως στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τον ταξιδιωτικό τομέα, θα πρέπει επίσης να ενημερώσουμε το κεκτημένο για το ψυχιακό έτος και είχαμε το 1990 κά κάτι αποφασίσει. Το, ο κόσμος όμως από τότε έχει αλλάξει. Οι συνήθειες ε, είναι διαφορετικές και χρειαζόμαστε να μπορούν οι καταναλωτές να αγοράζουν περισσότερα ταξίδια online, στο διαδίκτυο. Και εδώ θα πρέπει να προσαρμοστεί το κεκριμένο για τους ε, καταναλωτές στην ψηφιακή εποχή, εξυγχρονίζοντας το κεκριμένο όπου χρειάζεται ταυτόχρονα όμως βελτιώνοντας την επιβολή των ε, νόμων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, γιατί οι πολίτες έχουν το δικαίωμα σε αποτελεσματική και δίκαια δικαιοσύνη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε την εσωτερική αγορά στην οποία δρούν οι καταναλωτέ και η εσωτερική αγορά θα πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να προασπίσουν τα δικαιώματά τους. Ω ε, επίτροπο ε, δικαιοσύνη, υπεύθυνη για το θέμα αυτό, θέλω να εξασφαλίσω να είναι ε, η προστασία ίση είτε που αγοράζουν στις πατρίδες τους είτε αγοράζουν σε κάποια άλλη χώρα. Όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Ο ρόλος της Επιτροπής του Συστηματοφύλακα των Συνθήκων είναι να φροντίζει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν την νομοθεσία που έχουμε από κοινού υιοθετήσει. Θα πρέπει λοιπόν η επιβολή της νομοθεσίας αυτής να είναι ξεκάθαρη και ισότιμη σε όλα τα κράτη-μέλη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μάλκομ, η δική σας Επιτροπή γνωρίζει πάρα πολύ καλά την σημασία της ζωστής επιβολής του κεκτημένου μας και θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν θε, ε, θεωρεί πολύ σοβαρά το ρόλο του σε αυτό το νομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Πράγματι, είναι ένα συνεχές ε, θέμα που δουλεύουμε εδώ στην Επιτροπή μας και ξέρετε ότι κάνουμε και μελέτες για την οδηγία όσον αφορά τις εμπορικές πρακτικές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για αυτές τις αγωγικές σας παρατηρήσεις. Τώρα το λόγο έχει ο Τζον Ντάλι, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις δικές του προπτικές και μετά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Λίσμπεργκ πριν να αρχίσουμε και μπούμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Λίσμπεργκ, κύριε και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΙΜΚΟ, ιδιαίτερα εσένα Μάλκομ, που οργάνωσε από κοινού με την Επιτροπή την ε, ακρόαση αυτή για την ατζέντα των καταναλωτών. Είναι πολύ σημαντικό που η ακρόαση αυτή λαμβάνει χώρα εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή φυσικά και δουλεύει στον τομέα ε, των δικαιωμάτων ε, των καταναλωτών, αλλά έχει υποφεληθεί πάρα πολύ από το έργο της δικιάς σας Επιτροπής τη ΣΥΜΚΟ. Αυτό φαίνεται από τις πολυάριθμες εκθέσεις υψηλού επίπεδου που έχετε ετοιμάσει. Στις σημερινές συνθήκες όπου βρίσκεται η οικονομία μας, φυσικά και περιμένουμε με ανυπομονησία την έκθεση για τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους εισηγητές ε, της ΣΥΜΚΟ είναι εδώ και θα πάρουν το λόγο και τους είμαι ευγνώμων γι' αυτό, για τις εκθέσεις τους. Και μιλάω εκ μέρους όλων να σας πω ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συζήτηση, η οποία θα συνεισφέρει πάρα πολύ στην προετοιμασία Τη ατζέντα του καταναλωτή. Θα σας πω εγώ τώρα λιγάκι πώς βλέπω εγώ το μέλλον αυτή τη ατζέντα για τον καταναλωτή. Για μένα πρόκειται για ένα μέσο προκειμένου να πετύχουμε ένα σκοπό και ο σκοπός είναι να ενισχύσουμε με ένα όσο γίνεται καλύτερο πλαίσιο τον καταναλωτή. Γιατί ένας μημένος καταναλωτής δεν είναι μια απλή ιδέα, αποτελεί ένα πλαίσιο ιδεών και μηχανισμών προκειμένου πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές να μπορούν να ζήσουν μέσα σε μια βιώσιμη οικονομία και να συμμετέχουν σε αυτήν όλοι. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε τα μέσα για να μπορούν να αποφασίζουν εν γνώση των συνεπειών. Όπως αναγνωρίστηκε και πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η εμπιστοσύνη του καταναλωτή είναι και τα θεμέλια της ανάπτυξης. Και γι' αυτό και πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα όραμα για την πολιτική καταναλωτών μέσα στα επόμενα χρόνια. Για να πετύχουμε τους συνολικούς στόχους για το 2020, προκειμένου να έχουμε μία βιώσιμη ανάπτυξη στην οποία θα συμμετέχουν όλοι. Το μυστικό λοιπόν είναι ενίσχυση του καταναλωτή. Ο καταναλωτή να μπει στην καρδιά της ενιαία αγορά. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι ο καταναλωτή θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην εσωτερική αγορά. Να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα επιλογή και να ε, επιβάλλει και τα δικαιώματά του. Έτσι θα χτιστεί η εμπιστοσύνη. Έτσι λοιπόν ο καταναλωτής πρέπει να βρίσκεται, να αντιμετωπίζεται με δικαιοσύνη και επίσης όρις μέσα στον ανταγωνισμό. Χρειάζεται λοιπόν μια συνεκτική και συνολική αντιμετώπιση. Πολλά βέβαια έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για θέματα που παραδοσιακά συνδέονται με την πολιτική των καταναλωτών αλλά και σε διάφορους άλλους τομείς. Παρ' όλα αυτά, αν δεν υπάρχει συντονισμό, η αντιμετώπιση μας θα είναι κατακαιρματισμένη. Όσον αφορά τώρα την δομή της πρότασης, πιστεύω ότι η ατζέντα του καταναλωτή πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις πυλώνε που να καλύπτουν το σύνολο της σύγχρονης πολιτικής για τον καταναλωτή. Εννοείται ότι θα συζητήσουμε αυτούς τους πυλώνες αργότερα. Πρώτα απ' όλα, ασφάλεια. Όσον αφορά τα προϊόντα, τα αγαθά, τα τρόφιμα, αυτή είναι μια προϋπόθεση για οποιαδήποτε πολιτική καταναλωτή. Ασφάλεια, λοιπόν. Όταν αναθεωρηθεί η οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων, στόχος μας πρέπει να είναι να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο και η εποπτεία και επιθεώρηση ο έλεγχος να είναι πιο αποτελεσματικός. Γιατί υπάρχει και η παγκοσμιοποίηση, οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πώς θα λάβουμε καλύτερα υπόψη μας και την ασφάλεια και των υπηρεσιών. Δεύτερον, αν ε, θέλουμε ο καταναλωτής ε, να έχει περισσότερα δικαιώματα, πρέπει να μπορεί να έχει και πρόσβαση στην ενημέρωση και στις πληροφορίες. Η αγορά γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, άρα χρειάζεται η ενημέρωση να δίνεται με διαφάνεια και να είναι έγκυρη. Θα πρέπει όλη οι να είναι αξιόπιστοι και αντικειμενικοί. Σήμερα γίνονται προσπάθειες για ενημέρωση των φοιτητών, για παράδειγμα, οι οποίοι είναι οι καταναλωτέ του αύριο. Πρέπει λοιπόν να είναι ενημερωμένοι και να ξέρουν για να μπορούν να αποφασίζουν καλύτερα. Έπειτα, χρειάζεται αξιολόγηση τη δράση μα στον τομέα αυτό. Το θέμα τη εκπαίδευση, τη διαπαιδαγώγηση, τη κατάρτιση το λεβαίνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μα και θέλουμε μια διαδραστική πλατφόρμα για να συγκεντρώσουμε τι βέλτιστέ πρακτικέ. Οι οργανώσει των καταναλωτών επίση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο εδώ μπορούν να βοηθήσουν. Το προφίλ των οργανώσεων των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε να είναι περισσότερο ορατή και πρέπει η φωνή του καταναλωτή να είναι πιο δυνατή και να συμμετέχει στην εκπόνηση της πολιτικής. Χρειάζεται ενίσχυση των οργανώσεων καταναλωτών σε διάφορες χώρες μέλη. Έρχομαι στον τρίτο πυλώνα, διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε διάφορους τομείς πολιτικής. Για παράδειγμα, το βαθμολόγιο έχει δείξει ότι οι τραπεζικές μας ε, υπηρεσίες είναι προβληματικός τομέας για τους καταναλωτές. Έχουν γίνει προσπάθειες για αυτορύθμιση που όμως δεν ήταν επιτυχής. Γι' αυτό και θέλουμε να περάσουμε στα επόμενα βήματα. Η Vivian αναφέρθηκε σε διάφορα νομοθετικά, σε διάφορες νομοθετικές προσπάθειες που θα γίνουν. Τέταρτος πυλώνας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα τίθεται σε εφαρμογή το πλαίσιο που θα δημιουργήσουμε. Θα πρέπει χωρίς υψηλό κόστος ο καταναλωτής να μπορεί να προσφεύγει. Γρήγορα, εύκολα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με τις προτάσεις μας για τις εναλλακτικέ ε, μεθόδους διευθέτησης διαφορών. Με τις εθνικές αρχές πρέπει να συζητήσουμε για να ενισχυθούν τα δικαιώματα του καταναλωτή. Και όσοι ε, έμποροι δεν συμπεριφέρονται σωστά θα πρέπει να βγουν από την αγορά. Είναι πολύ βασικό οι εθνικές αρχές να επιβάλλουν τις διατάξεις για να προχωρήσουμε λοιπόν χρειάζεται ε, καλός συντονισμός μεταξύ μας, μεταξύ των δικτύων δικαιωμάτων καταναλωτών, μεταξύ κέντρων για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και διάφορες ε, νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εμπόριο για παράδειγμα, που έχει να κάνει με ε, βιώσιμες μορφές κατανάλωσης. Οι καταναλωτές θα πρέπει εύκολα να μπορούν να επιλέγουν. Δεν θα πρέπει να αποφασίζουμε, για παράδειγμα, για τα ε, απόβλητα χωρίς τη συμμετοχή των καταναλωτών. Όλα αυτά είναι βέβαια μια δύσκολη πρόκληση που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία σήμερα που βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση και βασιζόμαστε πάρα πολύ στην ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε και μια οριζόντια πολιτική καταναλωτών, αλλά σε διάφορους τομείς κλειδί όπου είναι ευάλωτος ο καταναλωτής, ε, αυτά να μην τα παραβλέψουμε. Θέλω επίσης να σας πω τελειώνοντα ότι για μένα η πολιτική για τον καταναλωτή είναι μια αναγκαιότητα που μας βοηθάει να έχουμε στη διάθεσή μα τα μέσα που χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε τον καταναλωτή και για να πετύχουμε μια καλή και βιώσιμη ανάπτυξη. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω πάλι τα περί ασφάλειας, κατάρτισης, διαπαιδαγώγησης, επανόρθωσης κλπ. Είμαι πεπισμένος ότι μια δυνατή πολιτική για τον καταναλωτή που να βασίζεται στα στοιχεία που σας έδωσα και μπορεί και θα αποτελέσει το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά. Οι καταναλωτές θα έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά και θα μπορέσουν έτσι να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη την οποία τόσο πολύ ανάγκη έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Τζον, γιατί παρουσίασε τα βασικά στοιχεία που θέλουμε να υπάρχουν σε μια ημερήσια διάταξη για τον καταναλωτή, καθώ και διότι έθεσε τους όρους για τις επόμενες ε, ε, τέτοιου είδους συναντήσεις. Να σας πω επίσης ότι μελέτησα και κάποια έγγραφα που δημοσιεύθηκαν χθε το βράδυ για, την, ε, για τον ευάλωτο χαρακτήρα του καταναλωτή. Ήταν μια ευτυχή σύμπτωση, αλλά να μιλήσουμε και στον παραπέμπω και στην εισηγήτρια που θα πάρει το λόγο αργότερα. Για να ολοκληρώσουμε τώρα με τις εισηγήσεις θα δώσω το λόγο στον πρέσβη της Δανίας και μετά θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε ερωτήσεις. Ανοίγω λοιπόν τώρα τον κατάλογο μιλητών για όσους είστε εδώ και αν έχουμε χρόνο θα ακούσουμε ίσως και ερωτήσεις από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Μπορείτε να ζητήσετε το λόγο, παρακαλώ. Λοιπόν, ε, κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Χάρμπορ και ευχαριστώ πολύ ε, το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάλεσαν την Δανική Προεδρία σε αυτήν την διάσκεψη καθώς και για τα θερμά σας ε, το θερμό σας καλώς όρισμα. Όντως, η Ιδανική Προεδρία αποδίδει μεγάλη προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη περί καταναλωτή κατά τη διάρκεια των έξι μηνών, όπου θα προεδρεύουμε των συζητήσεων εντός του Συμβουλίου. Το πρόγραμμα εργασίας μας για τους επόμενους έξι μήνες Ε, αποκαλείται η Ευρώπη στην δουλειά και μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές είναι η ασφαλής Ευρώπη και η δυναμική Ευρώπη. Πράγμα που νομίζω ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τα θέματα του καταναλωτή. Σίγουρα εμείς προσβλέπουμε, στον, προσμονούμε την ε, λήψη της στρατηγικής ε, μετά από την υφιστάμενη στρατηγική περί καταναλωτική, πολιτικής περί καταναλωτή που είναι μια καλή βάση για να βασιστούμε για τον, ε, τη στρατηγική μας δουλειά και τον προγραμματισμό μας σε συνεργασία με την Επιτροπή σας, την έκθεση Γκρέκ, Σάλτερ Μόζε για την ασφάλεια των προϊόντων και διάφορες εκθέσεις θα μπορούσα ακόμα να σας αναφέρω, που νομίζω θα εμπνεύσουν όχι μόνο την Κομισιόν στην δουλειά της σύνταξης της στρατηγικής για τον καταναλωτή, αλλά και το Συμβούλιο ε, που εργάζεται από αυτές τις βάσεις. Σε σχέση με τα σχόλια του Επιτρόπου Ντάλι, Θα ήθελα να τονίσω και να επικυρώσω ότι το Συμβούλιο επίσης πιστεύει πως οι βασικά κλειδιά, έννοιες κλειδιά, ε, θα πρέπει να είναι η χειραφέτηση των ε, καταναλωτών και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Αυτές οι λέξεις κλειδιά είναι στόχοι, αλλά είναι και μέσα. Μέσα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, και να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αλλά επίσης είναι και οι δείκτες για τον βαθμό στον οποίο έχουμε επιτύχει. Χρειαζόμαστε να έχουμε πληροφορίες για αυτές τις έννοιες, χρειάζεται να μπορούμε να τις μετρήσουμε για να αξιολογήσουμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τη σωστή πορεία. Δύο συγκεκριμένες προτεραιότητες θα ήθελα να τονίσω στην νομοθετική ατζέντα για την Δανική Προεδρία. Καταρχήν έχουμε το πρόγραμμα καταναλωτή και το δεύτερο είναι οι δίδυμες προτάσεις για εναλλακτική επίλυση διαφορών και για online επίλυση διαφορών. Καταρχήν το πρόγραμμα του καταναλωτή ε, εντάσσεται μέσα στο πολιετές ε, ε, πρόγραμμα, οπότε δεν μπορέσουμε να κλείσουμε το φάκελο αυτό μέσα στην Ιδανική Προεδρία, αλλά τουλάχιστον θα βρούμε, ελπίζουμε, μια συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη στους επόμενους 6 μήνες για αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Μπορεί να μην, ε, να μην είναι μεγάλα τα νούμερα σε σχέση με το γενικό πολιτέ πρόγραμμα, αλλά ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσει να συμβάλλει σε περισσότερη ενημέρωση, καλύτερη αίσθηση του πού ε, έγκυται η προκλήση ε, και χειραφέτηση της κοινωνίας των πολιτών και του καταναλωτή. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, στο οποίο θα δουλέψουμε για να έχουμε συμφωνία και στις μελλοντικέ προεδρίες με την Κυπριακή Κυβέρνηση που θα συνεργαστεί με το Ευρωκοινοβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας Και έπειτα έχουμε συγκεκριμένα νομοθετικά προγράμματα προς καλύτερη εφαρμογή, επιβολή της ε, ισχύωσης νομοθεσίας. Μια δυνατότητα είναι ε, οι προτάσεις περί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και online επίλυσης διαφορών. Δεν σημαίνει μόνο την αποκατάσταση και τη βελτίωση της επιβολής των δικαιωμάτων, αλλά νομίζω πως θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη και σημαντική συμβολή και γι' αυτό και είμαστε ευχαριστημένοι ότι, που βρίσκεται μέσα στα ένα, αποτελεί ένα από τα 12 ε, κλειδιά, δράσεις κλειδιά μέσα στο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Και έτσι οι κυβερνήσεις τόνισαν μόλις τέλη Ιανουαρίου ότι ελπίζουν πως αυτές οι προτάσεις θα μπορέσουν να αποτελέσουν πραγματικότητα, να μετατραπούν μάλλον σε, να υλοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο φέτος. Πολύ φιλόδοξο στόχο, αλλά με ευχαρίστηση μπορώ να σα πω, να σας πω ότι ήρθα σε επαφή με την κυρία Τούνον Χόνσταν και τον κύριο Γκρέχ, του συζητητέ, και έχω την εντύπωση πω είναι δυνατόν να δουλέψουμε σκληρά να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία και σίγουρα εμεί έχουμε την πρόθεση αυτό να το κάνουμε με τη βοήθεια τη επίτροπή. Και αυτά όλα είναι πολλά υποσχόμενα. Και αυτό γιατί, γιατί οι προτάσεις δεν βασίζονται, δεν, μάλλον δεν φτιάχνουν νέες ευρωπαϊκές δομές, αλλά βασίζονται στις υπάρχουσες δυνατότητες για τις εναλλακτικέ δυνατότητες επίλυσης διαφορών με εμπόρους και να τις επεκτείνουν όπου είναι αυτό δυνατό σε εθνικό επίπεδο και έτσι να εξαλείψουμε τις διαφορές που είχαμε στα, ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, και έτσι να μπορούμε να έχουμε μια κοινή πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Ε, να σας πω, να ολοκληρώσω λέγοντας ότι Έχουμε συγκεκριμένη δουλειά μπροστά μας, μαζί με τους δύο, συνομο... δύο συνομοθέτες μάλλον, χάρη στις πρωτοβουλίες της Κομισιόν. Οι προτάσεις δεν αφορούν μόνο τα δικαιώματα του καταναλωτή, αλλά και την εξασφάλιση της ανάπτυξης και την ε, χρήση, την αξιοποίηση ε, του πλήρους δυναμικού της ψηφιακής ενίας αγοράς και ως εξάμενη Προεδρία του Συμβουλίου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας δυναμικής και ασφαλούς Ευρώπης μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο επί τη βάση των προτάσεων της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Well, thank you uh, very much, uh, all Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις ομιλητές. Έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Και μετά έχουμε και άλλους ομιλητές. Καλή κυρία Ράπτη έχει πει ότι θέλει να υποβάλει κάποια ερώτηση, οπότε παρακαλώ, έχετε το λόγο. Και μετά έχουμε κατάλογο μιλητών, όποιος άλλος θέλει να πει. Όπως είπα και νωρίτερα, οι ενδιαφερόμενοι που βρίσκονται εδώ και θέλουν να παρέμβουν μπορούν να μας στείλουν ένα σημείωμα που να γράψουν το όνομά τους να ξέρουμε. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω τους δύο επιτρόπους και τους άλλους ομιλητές και τους ευχαριστώ που είναι εδώ για μια ακόμη φορά να μας ενημερώσουν. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να ακούσω την κυρία Ρέντινγκ από την αρχή. Ε, θέλω να, ε, να σας βάλω λιγάκι στο κλίμα πώς να πω, στη, στην σύνδεση αυτών που συζητούμε εδώ για τους καταναλωτές και στην πραγματική ζωή. Ε, προέρχομαι από την Ελλάδα, η οποία αργά τη νύχτα χθες, ξημερώματα σήμερα, έλαβε ε, αποφάσεις για πάρα πάρα πολύ σκληρά μέτρα λιτότητας. Η λιτότητα κάνει τους καταναλωτές περισσότερο συνειδητοποιημένους όταν έχεις λιγότερο χρήματα, λιγότερα χρήματα και τα καταναλώνεις, σκέφτεσαι διπλά πού καταναλώνεις αυτά τα χρήματα, τι προϊόν αγοράζεις και τι δικαιώματα έχεις στην περίπτωση που το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό. Έτσι λοιπόν να ε, ρωτώ ε, κυρίως τον Επίτροπο Νταλή, τον άκουσα να μιλάει για τον εναλλακτικό τρόπο για το ADR, το Alternative Dispute Resolution, αλλά δεν άκουσα, ίσως, ίσως κάνω λάθος, δεν άκουσα να κάνουμε κουβέντα για το collective redress. Και το collective redress που κατά τη γνώμη μου μειώνει το κόστος για τους καταναλωτές που πλήττονται ε, είναι ένα θέμα που υπάρχει πάντα στο Κοινοβούλιο, υπάρχει πάντα στους θεσμούς και θυμίζω ότι στην προηγούμενη Ολομέλεια ψηφίστηκε η έκθεση του κυρίου Λένε από την Επιτροπή Γιούρη. Ε, αυτό το θέμα ήθελα να θέσω υπόψη σας και να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη δουλειά που κάνετε και για την θετική σκέψη που έχετε για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Um, ναι, νομίζω ότι ο Επίτροπος ε, Ντάλι πρέπει να απαντήσει, αλλά ναι, και η Vivian ρέντινγκ. Όσον αφορά το EDR, γνωρίζετε ότι έχουμε αναλάβει τα πρώτα βήματα ήδη για να προχωρήσουμε για αυτό το θέμα και ε, με τους διαφορούς εταίρους και για τις διαδικασίες ADR προκειμένου να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, αν μη τι άλλο, κοινών προδιαγραφών. Μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο της κάθε χώρας μέλους. Ξέρετε ότι είναι ένα γιγάντιο έργο να καταφέρουμε να συμβάσουμε τις απόψεις των διάφορων χωρών, αλλά πιστεύω ότι προτείνεται ένα πολύ καλό σύστημα προκειμένου να έχουμε έναν κοινό παρονομαστή για το NDR και έτσι να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε στα εθνικά μας συστήματα. Ξέρετε, προχωράμε και την ψηφιακή ατζέντα, όπως είπε και η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ νωρίτερα. Η ψηφιακή αγορά είναι κάτι που θέλουμε επίσης να πιέσουμε. Και πιστεύουμε ότι αν αυξήσουμε την ψηφιακή αγορά από το μείον 5% όπως είπε η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ και φτάσουμε στο 15% του λιανικού εμπορίου, θα κερδίσουν οι καταναλωτές 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε λοιπόν για μεγάλα ποσά και για πολύ σημαντικά κίνητρα για μας. Βέβαια, ο καταναλωτής πρέπει να νιώθει εμπιστοσύνη. Άρα χρειάζεται μια διαδικασία διευκόλυνσης για τον καταναλωτή, προκειμένου αυτός να μπορεί πιο εύκολα να ακολουθήσει τη διαδικασία EDR σε οποιαδήποτε χώρα, γιατί θα είναι διασυνοριακό βέβαια το σύστημα, έτσι. Οπότε θα πρέπει να μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε χώρο που αγόρασαν τα αγαθά τους και να ζητήσουν ικανοποίηση εκεί. Προχωράμε για το θέμα των συλλογικών επανορθώσεων, συλλογικών προσφυγών. Προχωράμε με τον κύριο Αλμούνια και με την Βίβιαν βέβαια, η οποία θα μπορέσει να σας εξηγήσει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ναι, μετά τα όσα είπε ο συνάδελφος Ντάλι μόλις τώρα, πρέπει να προσθέσω ότι όντως οι εναλλακτικές ε, αυτές μέθοδοι επίλυσης διαφορών θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Η μελέτη που κάναμε έδειξε ότι χάνεται πάρα πολύ χρόνος όταν ε, δεν ζητάμε διαμεσολάβηση. Κάπου 400 επιπλέον μέρες χάνονται. Κάπου 13.000 ευρώ για κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλό που ο συνάδελφος ε, Νταλή θέτει ε, τα θέματα αυτά επιτάπητος. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι έχουμε και μία οδηγία ε, διαμεσολάβησης. Η οδηγία αυτή θα πρέπει ήδη να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες μέλη. Εφόσον 21 Μαΐου 2011 καταλήξαμε. Άρα λοιπόν τώρα εξετάζουμε πώς έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Και έχω διαπιστώσει ότι σε ορισμένες χώρες οι κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την οδηγία όχι μόνο για διασυνοριακές περιπτώσεις, αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο, μέσα στην ίδια τη χώρα. Κάτι που είναι ιδιαίτερα θετικό. Σε ορισμένες χώρες χρησιμοποίησαν την διαμεσολάβηση ως υποχρεωτικό μέσο, βέβαια εξαρτάται από την φύση της διένεξης ή από τα οικονομικά κίνητρα και κυρώσεις, άλλοι πάλι το χρησιμοποιούν και στο εσωτερικό και διασυνοριακά. Πέντε χώρες μέλη μέχρι τώρα δεν έχουν κοινοποίησει ότι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας για να ξεκινήσει μια διαδικασία επί ε, προσπαθούμε να πιέσουμε τις χώρες να κάνουν τη δουλειά τους πρώτα απ' όλα. Γιατί στόχος μας δεν είναι βέβαια να πάμε μια χώρα στο δικαστήριο. Στόχος μας είναι, όπως και με τη διαμεσολάβηση, όπως προτείνει και αυτή, να λύνονται τα προβλήματα πριν φτάσουμε στα δικαστήρια. Ελπίζω λοιπόν να το καταφέρουμε αυτό. Και έχω δει ότι πέντε χώρες που λείπουν, που δεν το έχουν κάνει ακόμα, ε, κάπως ξεκινάνε. Για τις συλλογικές προσφυγές τώρα. Υπάρχουν τρεις επίτροποι, όπως είπε και ο Τζον πριν από λίγο, Αλμούνια, Ντάλι και Ρέντινγκ. Και οι τρεις λοιπόν συνεργαζόμαστε για να προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Πήραμε επιστολή από τον πρόεδρο Λένε, ο οποίος ζητάει από τον πρόεδρο Μπαρόσο να καθυστερήσουμε λίγο, να περιμένουμε να αποφανθεί το κοινοβούλιο πρώτα. Ε, τώρα αποφάνθηκε το κοινοβούλιο. Οπότε εννοείται ότι λαμβάνουμε υπόψη μα τα όσα είπε το Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήτανε. Ή πριν από δύο, δεν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει έχουμε τώρα ε, τα στοιχεία <coughs> αυτά. Ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το δικό μας το έργο. Εσείς λέτε ως Ευρωβουλευτής ότι θέλετε οριζόντια ε, μέσα. Το πήραμε το μήνυμα. Οι τρεις επίτροποι θα προχωρήσουν σε βάθος για τη δουλειά τους και πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Το πρόγραμμα εργασίας πάντως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012 προβλέπει δράση για τις συλλογικές προσφυγές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι λοιπόν που μπορέσαμε έτσι και απαντήσαμε. Θα ζητήσω από τους συναδέλφους μικρά σχόλια, εφόσον έχουν, ο κύριος Τρενταφυλλίδη σε λίγο, σε λίγο, μια στιγμή. Να σας πω ποιος είναι ο κατάλογος ομιλητών για να κάνετε σύντομες παρακαλώ ερωτήσεις. Έτσι. Και οι προσκεκλημένοι μας θα μπορέσουν να μιλήσουν. Um, be... και Σβάμπε πρώτα απ' όλα για ερωτήσεις. Και μετέχουμε έχουμε την κυρία Ευαγγελία Κακελάκη. Συγγνώμη αν ε, δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Ξέρω ότι είσαστε Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή παρατηρητής και μετέχουμε έχουμε τον κύριο Χάντριξεφ από την Σουηδική Οργάνωση Καταναλωτών και Καρέλη επίσης από την Ιταλία, από την Οργάνωση Καταναλωτών εκεί. Θα σας δώσω το λόγο για σύντομες ερωτήσεις. Έτσι, Τριανταφυλλίδης πρώτα όμως. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές ε, και την Επιτροπή που υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών και γιατί ο καταναλωτής πρέπει να είναι πιο ισχυρός ενισχύοντας τα δικαιώματά του και τις δυνατότητες που έχει πρόσβασης ε, σε επίλυση διαφορών. Η ερώτησή μου είναι για την νομοθεσία. Ένα νέο πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020, νέα ατζέντα για το 2015-2020. Αναρωτιέμαι, είναι αναγκαία όλα αυτά ή μήπως θα μπορούσε να υπάρχει συντονισμός έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα τα πράγματα και για μας αλλά και για τον κόσμο. ΣΦΑΠ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατεχήν θέλω να ευχαριστήσω τα όσα μας είπε η κυρία Αντιπρόεδρε ε, Ρέντινγκ χθες ε, στη Βουλγαρία και η Ρουμανία είδαμε ότι δεν λειτουργεί επαρκώς η δικαιοσύνη στις χώρες αυτές. Και νομίζω ότι εκεί όταν αναλύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το θέμα της δικαιοσύνης. Γιατί τα δικαιώματα των καταναλωτών έχουν νόημα μονάχα αν μπορούν να επιβληθούν. Ποια είναι η εκτίμησή σας για την επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν τη σωστή μέθοδο δικαιοσύνης ακόμα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχω μία ερώτηση για την ε, κυρία Ρέντινγκ. Ε, αναφέρατε στην ε, τοποθέτησή σας ότι η ε, καινούργια πρόταση της Επιτροπής για την ε, κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πωλήσει προβλέπει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ε, καταναλωτών. Ε, έχετε υπόψη σας ότι σε αρκετά κράτη-μέλη αυτή η προστασία υποβαθμίζεται και είναι αναγκασμένα αυτά τα κράτη-μέλη να μειώσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών για να μπορέσει να εφαρμοστεί η μέγιστη εναρμόνιση με αυτή την πρόταση, σύμφωνα με αυτή την πρόταση της Επιτροπής. Προέρχομαι από την Ελλάδα και έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα και όσον αφορά τις εγγυήσει για τα ελαττωματικά προϊόντα και όσον αφορά τους ε, καταχρηστικούς όρους της συμβάσης. Θα υποχρεωθεί η Ελλάδα να υποβαθμίσει την ομοθεσία της. Θα ήθελα να ξέρω αν είστε γνώστης αυτού του προβλήματος και τι προτίθεστε να κάνετε. Ευχαριστώ. Good, thank you very much. Um, Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Thank you for this opportunity. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που αφορά και τους δύο επιτρόπους όσον αφορά την παρουσία των θαυμασίων πρωτοβουλειών που παρουσιάστηκαν σε παραδοσιακούς τομείς της εργασίας όπου η Κομισιόν ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική και θα συνεχίσει να είναι αποτελεσματική. Υπάρχουν όμως νέες προκλήσεις στον κόσμο όσον αφορά την αηφόρο κατανάλωση και ελπίζω να μου πείτε και οι δύο επίτροπε πώς θα ενσωματώσετε αυτό το θέμα της εφόρου κατανάλωσης στη νέα ατζέντα για το καταναλωτή. Γιατί νομίζω ότι με τις προκλήσεις που έχουν μπροστά μας όσον αφορά την οικονομία και το περιβάλλον πρέπει να έχουμε μια πολιτική καταναλωτών που θα αναφέρεται και σε αυτό το θέμα αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λεπρός, πολύ ωραίες ερωτήσεις. Σικαρέλη, buongiorno, grazie per questa occasione di confronto. Io volevo sottolineare intanto... Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε εδώ να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιε ερωτήσει. Υποστηρίζουμε βέβαια την ατζέντα για το καταναλωτή και την άμεση συμμετοχή τους. Σημαντικό. Η ερώτηση μου είναι εξή. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις δράσεις που προτίθεστε να αναλάβετε για να υποστηρίξετε τα δικαιώματα των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά το θέμα του συστήματος δικαιοσύνης. Προβλέπετε κάτι ώστε να είναι πιο εύκολα ενός των καταναλωτών να προσφύγουν στα δικαστήρια. Συλλογικές δηλαδή προσφύγες Προβλέπετε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό θα δώσει δυνατότητα σε άτομα που δεν έχουν τους πόρους να μπορούν να προσφύγουν παρόλα αυτά στη δικαιοσύνη για θέματα προστασίας του καταναλωτή. Τέλος, ποιες είναι οι δραστηριότητες που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά σας για να βοηθήσουν να μάθουν οι καταναλωτές πώς μπορούν να προστατευτούν. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε ίσως ε, ε, λίγο να έχουμε τις απαντήσεις στα θέματα αυτά. Ο Τζον Νταλή πρώτος. Θα ήθελα να σας κάποια τα θέματα που εθίγησαν. Καταρχήν ο το Πρωτοβουλίας και τα προγράμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή βέβαια μέσα στα πλαίσια του συστήματος που έχουμε στην Ευρώπη θα πρέπει να εξετάζουμε συγκεκριμένες πράξεις. Όταν αναφερόμαστε σε ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές, αναφερόμαστε καταρχήν στο οικονομικό πλαίσιο και μετά θα πρέπει να προσθεθούν οι διάφορες δράσεις για τους καταναλωτές. για να έχουμε τους απαραίτητους πόρους και τις δομές και τη νομική βάση για να μπορέσουν να λεφθούν οι δράσεις αυτές, Για επιτευχθούν οι στόχοι μα. Uh, Γιατί καμιά φορά, γι' αυτό καμιά φορά υπάρχει κάποια σύγχυση με τους διάφορους όρους και μέσα και όργανα που ε, χρησιμοποιούμε. Και εγώ το μαθαίνω σιγά σιγά. Πρέπει να τα ετοιμάσουμε όλα αυτά για να μπορούν να ληφθούν οι δράσεις. Αηφορία. Κάτι που έθιξε και η κυρία Ράπτη. Και εσείς τώρα. Ιδίως αυτή την κατάσταση τώρα της, των μέτρων λιτότητας υπάρχει έντονη κοινωνική πίεση στους πληθυσμούς. Και νομίζω ότι ε, οι κατανοητές είναι όσο πάει και περισσότερο σημαντική, ζωτική θα έλεγα και μπορούν έτσι να είμαστε σίγουροι ότι οι κατανοητές έχουν όλα τα μέσα στα χέρια τους που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν αηφόρο ε, όχι μόνο για το περιβάλλον για να μειωθούν τα απόλυτα κλπ. αλλά και όσον αφορά τον προπολογισμό. Πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Πρέπει να μην ξεπερνάμε δηλαδή τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας στην καθημερινή μας ζωή και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές, ε, να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις στην αγορά όταν αποφασίζουμε τι θα ψωνίσουμε, τι θα αγοράσουμε. Και θα πρέπει έτσι να συνεχίσουμε να πιέσουμε και να εκπαιδεύουμε τους καταναλωτές για το πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν και βλέπετε ότι παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις για την, ε, για την ετικετοθεσία, για τη σήμανση, για όλα αυτά, για τα προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τον καταναλωτή πώς θα μπορεί να ερμηνεύει και να χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες αυτές που του δίνουμε με τον καλύτερο ιδανικό τρόπο. Για το δική του προσωπικά, τις προσωπικές ανάγκες. Μπορεί αυτό διαφέρει δηλαδή από τον καταναλωτή στον άλλο. Με τη βοήθειά σας βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε να συνεχίσουμε στη διακατεύθυνση. Όσον αφορά τις οργανώσεις των καταναλωτών, προσπαθούμε κι εμείς να αυξήσουμε το δυναμικό των οργανώσεων των καταναλωτών στα διάφορα κρατημέλη. Καταλαβαίνω, γιατί επισκέφθηκα με διάφορα κρατημέλη και μίλησα με διάφορους οργανώσεις των καταναλωτών, ότι υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες, ικανότητες, ε, υποστήριξη που έχουν αυτές οι οργανώσεις των καταναλωτών και άρα πρέπει να δράσουμε περισσότερο σε ορισμένα κρατημένα από τι άλλες για να είμαστε σίγουροι ότι οι καταναλωτές ε, έχουν τις δυνατότητες αυτές στις χώρες τους. Παραδείγματος άλλο το θέμα της ε, προσφυγής στη δικαιοσύνη ε, είναι κάτι που το εξετάζουμε. Πώς θα μπορεί να γίνει εκεί μια συμμετοχή των οργανώσεων των καταναλωτών. Θα μπορούσε να υπάρχει σωστή πίεση στο να δώσουμε περισσότερη ισχύ στις οργανώσεις των καταναλωτών και ε, επισκέφτηκα χώρες όπου γίνεται ήδη. Εκεί μπορούμε νομίζω να προσπαθήσουμε και να πιέσουμε. Οι ιδιωτικέ οργανώσει, μη κυβερνητικέ οργανώσει στι διάφορε χώρε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ για να δώσουμε όχι μόνο την σωστή εποπτεία της κατάστασης επιτόπου, αλλά να έχουν τα κράτη-μέλη και εμείς, όλοι δηλαδή που προετοιμάζουμε την νομοθεσία, να έχουμε τα επαρκή στοιχεία στα χέρια μας για να μπορέσουμε να βασίσουμε σωστά τις αποφάσεις μας. Ευχαριστώ. Well, you might not know me so well in this committee here as in other committees. Ίσως δεν είμαι εδώ τόσο γνωστή ότι, όσο σε άλλοι σε επιτροπές, αλλά εγώ είμαι ο τύπος του επιτρόπου που δεν θέλει να υπάρχουν πολλές εκθέσεις, αλλά θέλει κάτι συγκεκριμένο, νομοθεσία δηλαδή, νομοθετικές πράξεις. Πού το κρέας λέω. Έχουμε ένα πρόβλημα, ποια είναι η λύση του. Τούτου λεχθέντος υπάρχουν δύο ερωτήσει ερωτήσεις για τη δικαιοσύνη. Είναι αληθές. Αν κανένας, οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ένα σύστημα δικαιοσύνης που δεν λειτουργεί, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι και η οικονομία δεν λειτουργεί. Γιατί δεν υπάρχει πιστοσύνη για τους επενδυτές και δεν υπάρχει πιστοσύνη των καταναλωτών επίσης. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο σε όλα τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουμε και εξετάζουμε αυτά τα συστήματα δικαιοσύνης που έχουν ελλείψεις περισσότερο και το είπε ξεκάθαρο και ο Σβάπ. Έχουμε ορισμένα κράτη-μέλη όπου τα, ε, η, δικαιοσύνη είναι υπό επιτήρηση, Βουλγαρία και Ρουμανία συγκεκριμένα, αλλά και κάτι άλλο που ίσως δεν γνωρίζετε. Στις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πολύ έντονη οικονομική κρίση έχουμε δώσει τη δυνατότητα εμπειρογνώμονες δικαιοσύνη να ξαναδημιουργήσουν εκεί τη δικαιοσύνη. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα, όπως επίσης στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Και τώρα αρχίσαμε να στέλνουμε τους εμπειρογνώμονες και στην Ιταλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή το αστικό δίκαιο να λειτουργεί. Αν δεν λειτουργεί το αστικό δίκαιο, δεν υπάρχει καμία νομική, αβε, ε, νομική βεβαιότητα στις κοινωνίες μας. Αυτό είναι κάτι που δεν ακούγεται πολύ, αλλά γίνεται πάντως. Ε, τώρα, μία πληροφορία που δεν έχετε ακόμα ίσως δει. για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα ε, οργανώσεις των καταναλωτών να προσφύγουν στο δικαστήριο εξ ονόματος των καταναλωτών. Αυτό προβλέπεται στη νέα οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πάλι, όχι έκθεση, αλλά κάτι το συγκεκριμένο τα δικαιώματα δηλαδή των οργανώσεων των καταναλωτών, να βοηθήσουν τους καταναλωτές να βρουν το δικαιό τους. Ένα άλλο πρόβλημα για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων. Άκουσα τόσες εσφαλμένες δηλώσεις και εσφαλμένες ενημερώσεις όσον αφορά αυτή την νομοθετική πράξη. Και αν είχε δίκιο κύριε Κακυλάκη, θα ήταν πραγματικά πολύ κακή νομοθεσία αυτή. Ευτυχώς όμως δεν έχει δίκιο. Αυτός ο κατονομισμός δεν άπτεται των εθνικών κανόνων καταρχήν. Είναι μόνο για διασυνοριακές δραστηριότητες, ρητά. Και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί μόνο το 6% των καταναλωτών τολμούν να περάσουν τα σύνορα, γιατί φοβούνται ποια θα είναι τα δικαιώματά τους στην γειτονική χώρα. Δεν το ξέρουν. Δεν τους υποχρεώνουμε λοιπόν να επιλέξουν ένα καινούριο σύστημα, αλλά τους δίνουμε την δυνατότητα επιλογής, εάν το θέλουν. Και αυτό μόνο για αγορές διασυνοριακά. του λεχθέντος, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών έχει εισαχθεί ένα προς ένα στο νέο κανονισμό. Αλλά η οδηγία αυτή για τα δικαιώματα των καταναλωτών αφορά μόνο τρία σημεία από τα 18 του νέου κανονισμού. Ο νέος κανονισμός δηλαδή προχωράει πολύ περισσότερο, δίνει πολύ περισσότερα δικαιώματα από τη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Παραδείγματος όσον αφορά το θέμα της ε, διόρθωσης για ελαττωματικά προϊόντα και το δικαίωμα των καταναλωτών να θέσουν λήξη, να καταγγείλουν μια σύμβαση που έχουν υπογράψει. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάζετε αυτό που υπάρχει επιτάπητος και όχι να ακούτε μόνο αυτά που λέγονται σε κάποια ανακοινοθέντα. for δεν έχουμε χρόνο για παραπάνω ερωτήσεις, παρόλο που έχουμε άλλες τρεις εδώ. Δεν ε, ακούγεται ο μιλήτρια εκτός μικροφώνου. Συγγνώμη, αλλά η κυρία Ρέντιν, και μιλάω για προσωπικό θέμα, ε, μελέτησα την πρόταση. Την μελέτησα. Και υπάρχουν κάποιοι όροι που λένε ότι τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν αυτό το θελοντικό μέσο στην εθνική τους νομοθεσία. Αυτό είναι ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όταν ο καταναλωτής δέχεται αυτό το θελοντική βάση μέσο, δεν ε, μπορεί να επωφεληθεί από το ροουμένα. από τη Ρώμη 1. Δεν μπορεί. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι είναι επίμαχο το θέμα. Υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα και χρειαζόμαστε διευκρινήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Very quickly. First... Πολύ σύντομα να σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, προκειμένου να είμαστε όλοι ήρεμοι για αυτό το θέμα. Η Επιτροπή Τζουρί η Νομική Επιτροπή, θα οργανώσει τέσσερις δημόσιες ακροάσεις για τα διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το common sense law. Με δύο λόγια δηλαδή, το ένα είναι σωστό, όπως και στη περίπτωση αυτή για τις περισσότερες χώρες μέλη αυτό τι θα σημαίνει. Θα σημαίνει επιπλέον δικαιώματα από αυτά τα οποία έχουμε σήμερα. Για το δεύτερο δεν είναι αλήθεια. Δεν αλλάζει το Rome 1 με την νομοθεσία αυτή. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τόσο ζωντανή ανταλλαγή ερωτήσεων-απαντήσεων. Έχουμε και τρεις ακόμα ομιλητές. Παραμένει το όνομά του στον κατάλογο ομιλητών. Πάντως ε, θέλω να ευχαριστήσω τους επιτρόπους και τους δύο για την παρουσία τους εδώ που μας έκαναν τις παρουσιάσεις τους στην αρχή και απάντησαν στη συνέχεια στις ερωτήσεις μας. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί τους και θα συνεχίσουμε εμείς τη συζήτηση για κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και θα θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουμε όλοι να δουλέψουμε για να βελτιώσουμε ολόκληρο το χώρο τη ενίσχυσης των δικαιωμάτων του καταναλωτή και την επιβολή της νομοθεσίας. Θα συνεχίσουμε όλα τα επόμενα χρόνια βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο με χειροκρότημα σας ευχαριστούμε. And if you give us a moment, we're just going to rearrange the Και σε ετοιμάσουμε εδώ το Προεδρείο για το επόμενο κομμάτι. so, ladies and gentlemen, can we now, um, can I invite you to um, resume your place? Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε την επόμενη, το επόμενο κομμάτι της συνεδρίασης. Can we have some, uh, Mr. Schwab and Mrs. Uh, Ruler, please? Uh, if we could uh, resume, thank you very much. Κύριε Σβάμπ, παρακαλώ καθίστε για να συνεχίσουμε. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Και εδώ θα ήθελα θερμά να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους ομιλητές που θα κάθονται εδώ από δεξιά. Δεν θα σας κατονομάσω χωριστά. Είμαι ευτυχής που δεν χρειάζεται να λέω ονόματα όλη την ημέρα. Έχω όμως ε, κάποιους ε, πολύ καλούς ε, εισηγητές εδώ. Έχουμε και έχουμε την κυρία Πάολα το story Κότζι, την Γενική Διευθύντρια και εγώ έτσι θα, δεν θα κάνω τίποτα για την υπόλοιπη συνεδρίαση. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Πάολα Τεστόρη Κότζη που είναι Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης για την Υγεία και τον, τους καταναλωτές και πριν το κάνω αυτό να σας πω ότι είμαι ευτυχής που είχαμε έτσι δυναμικές παρεμβάσεις από τους διάφορους ακροατές. Επίσης θα ήθελα να πω ποιους έχω στον κατάλογο μου. Which? Right, Ναι, σας εντόπισα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιοι είστε οι επόμενοι στον κατάλογο, αν θέλετε να παρέμβετε. Dano from uh, the Consumer Organization in Italy. Ο κύριος Πιέτρο Τζορτάνο από μια Ένωση Καταναλωτών της Ιταλίας. Α, εκεί βρίσκεστε. Ωραία, ευχαριστώ. Κορνίλια Τάους από την Γερμανική Ένωση Καταναλωτών. Είστε εδώ στον καταλογό μου. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο, σηκώστε το χέρι σας. Και Όποιο άλλο θέλει να μας στείλει την κάρτα του ή να μας στείλει ένα χαρτάκι μέσω των ε, κλητήρων, θα σας ε, βάλουμε στον κατάλογο μαζί με του συναδέλφους από το Ευρωκοινοβούλιο. Οι οποίοι θα έχουν την προτεραιότητα, αλλά τώρα που είδαν πόσο ποιοτική είναι η υπόλοιπη παρεμβαίνοντες από τους διάφορους οργανισμούς, θα πρέπει και εκείνοι να βάλουν τα δυνατά τους. Θα δώσω δε το λόγο πρώτα στον κύριο Τρενταφυλλίδη, γιατί όπως ξέρετε έχουμε κάνει σημαντική δουλειά για την ε, ατζέντα των καταναλωτών. Έχει πέντε λεπτά maximum για να μας παρουσιάσει την εργασία του. Κυριάκο, έχεις το λόγο λοιπόν. Ε, γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει γύρω στον μαιο Ιούνιο φέτος τη νέα πράξη για τα δικαιώματα των καταναλωτών που αφορούν την αναθεώρηση της πολιτικής για τους καταναλωτές, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Εσωτερική Αγορά, η Επιτροπή μας δηλαδή, συνέταξε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών. Τη σύνταξη της έκθεσης προηγήθηκε ανταλλαγή απόψεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδιαίτερα με τους συνδέσμους καταναλωτών και τους ίδιους του καταναλωτέ, με στόχο να ακουστούν οι προβληματισμοί τους, ώστε να επιτευχθεί και ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης που είναι η επανατοποθέτηση των καταναλωτών στην καρδιά της ενιαίας αγοράς δομημένη σε πιο γερές βάσεις την κοινωνικότητα και την βιωσιμότητα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να μεγεθύνεται και να εμβαθύνεται, θα πρέπει παράλληλα να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα επιτυχάνεται σε βάρος των εργαζομένων, των καταναλωτών γενικότερα και του περιβάλλοντος. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να προστατεύουν την υγεία και την ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας την καθιέρωση πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και αποτελεσματικότερους τρόπους αγοράς και κατανάλωσης των τροφών, προκειμένου να προλαμβάνεται και να καταπολεμάται η κατασπατάληση των τροφών. Πέραν τούτου, η νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στόχους για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ότι ο Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να είναι το επίκεντρο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη μεγέθυνση, καθώς και ότι σήμερα το 16,3% του πληθυσμού της Ευρώπης κινδυνεύει από φτώχεια. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι με τον τρόπο που συντελείται η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ο καταναλωτής έχει πάψει να την κρίζεται ως πολίτης και τίνει να αντιμετωπίζεται περισσότερο ως πελάτης. Οι καταναλωτές δεν συνιστούν μια ομοιογενή ομάδα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τις καταναλωτικές τους δεξιότητες και τη γνώση της νομοθεσίας. Σε μια ευρωπαϊκή κοινή αγορά των 495 εκατομμυρίων, παρατηρούνται διαφορετικές συνθήκες και ανισότητες που η έκθεση στοχεύει να μειώσει μέσα από την επανατοποθέτηση των καταναλωτών. Άρα, άμεσος στόχος της έκθεσης είναι προτάσεις για εξίσωση και αύξηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και καλύτερη ενημέρωση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την επίτευξη υψηλού επίπεδου προστασίας και ενδυνάμωσης του καταναλωτή με αποτελεσματική δημόσια εποπτεία της αγορά και επιβολή του νόμου. Γι' αυτό τον λόγο η έκθεση περιλαμβάνει ξεχωριστό κεφάλαιο με σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Θα πρέπει, για παράδειγμα, δεδομένης της αλματόδους αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ρυθμίσεις διασυνοριακών διαδικτυακών συναλλαγών, εκφράζεται δε η ανησυχία για το ότι η τρέχουσα έλλειψη αποζημίωση συνιστά σημαντικότατο κενό του νομικού συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον πίνακα αποτελεσμάτων του καταναλωτή το 44% των καταναλωτών δήλωσε αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώματα τους σχετικά με τις διασυνοριακές αγορές. Πρέπει λοιπόν να παρέχεται στους καταναλωτές και στους εμπόρους διαφανέστερη πληροφόρηση μέσω των κανόνων ενιαίας παρουσίασης των τιμών και ιστότοπων ακριβούς και διαφανούς σύγκρισης των τιμών στο διαδικτυακό εμπόριο. Πρέπει παράλληλα οι καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλίζεται ότι γίνονται πλήρως σεβαστά, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και ο ιδιωτικός τους βίος. Η προστασία του καταναλωτή θα εξασφαλιστεί μέσω της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά και μέσω της προσβασιμότητας σε αυτά. Είναι αναγκαίο λοιπόν να παρασχεθεί μεγαλύτερη ασφάλεια στα προϊόντα με μεγαλύτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι που εκ της φύσης τους είναι πολύ πιο ευάλωτοι με σχεδιασμό πολιτικών για τον καταναλωτή που θα λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ευάλωτων ομάδων, μείωση της έκθεσης των καταναλωτών σε επικίνδυνα προϊόντα και προστασία των παιδιών από την παραπλανητική διαφήμιση. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας και πρόσβασης σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι προδιαγραφές προκειμένου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να καταστούν προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές ανεξαρτήτως ηλικίας και σωματικών ικανοτήτων. Τέλος, παρατηρείται δυσαρέσκεια των καταναλωτών προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η οποία προέρχεται εν μέρει από τις κακές συμβουλές που λαμβάνουν. Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων των αγορών, η πλειονότητα των καταναλωτών δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τονίζεται δε η σημασία που έχει για τους καταναλωτές η διαφάνεια στις τραπεζικές χρεώσεις. Καταληκτικά, είναι πρωταρχική σημασία να εξασφαλιστεί εμπιστοσύνη, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στις συναλλαγές και εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας των καταναλωτών με ενεργή και ενιαία εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων μέσα από τον συντονισμό και την ενίσχυση των δράσεων εποπτείας της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ που έτσι είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε αυτή την πολύ σημαντική δουλειά. Και τώρα θα ακούσουμε την Πάολα Τεστόρη Κότζη. Σε αυτή τη συνεδρία θα μιλήσουμε για ασφάλεια των καταναλωτών. Ε, είναι η ασφάλεια η βάση οποιασδήποτε πολιτικής για τον καταναλωτή. Ασφάλεια τροφίμων, ασφάλεια υπηρεσιών. Τώρα εμείς ε, φέτος παρουσιάσαμε την αναθεώρηση, την Γενική Οδηγία περί ασφάλειας των προϊόντων, όπου εξετάζουμε και το θέμα της εποπτείας της αγοράς, που είναι θεμελιώδες θέμα, γιατί, γιατί δεν αρκεί να έχει κανείς κανόνες, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή τους και τον έλεγχο. Στη σημερινή συζήτηση λοιπόν θα δούμε εάν υπάρχουν σημαντικά θέματα τα οποία ε, να αφορούν την εποπτεία της αγοράς. Επίσης θα πρέπει να πω πως έχουμε εξεζήλευτο ρεκόρ γιατί είμαστε μια από τις καλύτερες περιοχές του κόσμου όσον αφορά τις απαιτήσει και τους ελέγχους αλλά κάποιες φορές φυσικά υπάρχουν ατυχήματα, συμβαίνουν ατυχήματα και αναθεωρούμε τις ε, ε, διατάξεις μας. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο καταρχήν στην κυρία Κριστέλ Σκάλντερμος από την DG IMCO που είναι η συγγήτρια για την αναθεώρηση της οδηγίας, της γενικής οδηγίας, μια έκθεση όπου σαφώς ε, μελετούμε την αποτελεσματικότητα για να λάβουμε υπόψη την θέση του Κοινοβουλίου. Κριστέλ λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα έλεγα ότι Πιστεύω πως αυτή η ακρόαση είναι πάρα πολύ σημαντική για να γνωρίζουμε σε ποιους τομείς θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας περισσότερο στο μέλλον όταν, όσον αφορά την ε, εσωτερική αγορά. Αλλά εγώ τον τελευταίο καιρό εστίασα την προσοχή στην ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Ε, εργάστηκα για το πακέτο περιτροφίμων πριν από κάποια χρόνια και ήμουν και εισηγήτρια εδώ στην ΙΜΚΟ όσον αφορά την, ε, την αναθεώρηση της, οδηγίας, της γενικής οδηγίας περί ασφάλειας των τροφίμων. Θα ξεκινούσα λέγοντας το εξής. Η ασφάλεια για τους καταναλωτές δεν είναι θέμα ε, προαιρετικό, πρέπει να είναι υποχρεωτικό ώστε να είναι ασφαλή, σίγουρα ασφαλή τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα συμβαίνει αυτό. Εδώ στο Κοινοβούλιο προτείναμε να γίνει μια γρήγορη αναθεώρηση γιατί έτσι θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε την νομοθεσία. Όμως για μένα οδηγία, γενική οδηγία για τα ενασφάλεια των προϊόντων δεν είναι το μόνο μέσο που έχουμε και πρέπει να αναθεωρήσουμε. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ και θέλω αυτό να το τονίσω για την λυπή εποπτεία της ενιαίας αγοράς σήμερα, διότι πιστεύω πως η νομοθεσία δεν είναι πολύ κακή. Έχουμε βελτιώσει την νομοθεσία, όμως βλέπουμε πως τα κράτη-μέλη δεν επιβάλλουν την ισχύουσα νομοθεσία με το σωστό τρόπο όχι αρκετά και όχι αρκετά γρήγορα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό για μένα, γιατί αν δεν έχουμε σωστή εποπτεία της αγοράς, τότε ο κόσμος που, κάνει απάτης με τα προϊόντα ε, ξεφεύγει. Και αυτό φυσικά βλάπτει τους καταναλωτές. Δεν αρκεί λοιπόν, χρειάζεται καλύτερη εποπτεία έτσι ώστε ε, οι καταναλωτές να εμπιστεύονται τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά μας. Αυτό θα πρέπει η κατάσταση να βελτιωθεί και ξέρω πως αυτός ο τομέας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο πιστεύω πως όταν μιλάμε για τους καταναλωτές και το πρόγραμμα για τους καταναλωτές για τα επόμενα χρόνια πρέπει κάτι να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Θα μπορούσε αυτό να γίνει μέσω νομοθεσίας, μέσω καλύτερου συντονισμού, καλύτερης χρήσης των πόρων, αλλά Πάντω σίγουρα θα πρέπει να πιεστούν περισσότερο τα κράτη-μέλη τα οποία δεν κάνουν αρκετά. Ορισμένε φορέ πιστεύω θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία όπου name and shame, όπου δηλαδή καταδεικνύουμε και δακτυλοδείχνουμε ε, τους δράστες. Ε, η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική, πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να βελτιώσουμε την νομοθεσία, αλλά σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε την εποπτεία και την επιβολή. Καλό λοιπόν την Κομισιόν και του συναδέλφου εδώ στο Κοινοβούλιο να κάνουμε κάτι σε αυτό το τομέα. Και σε εσά κάνω έκκληση, κύριε Πίτροπε. Ξέρω πω σα ενδιαφέρει το θέμα, ξέρω πω ανησυχείτε κι εσεί. Α ενώσουμε λοιπόν τι δυνάμει μα και α κάνουμε κάτι με τα κράτη-μέλη που δεν ε, ε κάνουν αρκετά. Γιατί στο κάτω-κάτω τη γραφή είναι θέμα εμπιστοσύνη και ασφάλεια των καταναλωτών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ισχυρότεροι. Αυτό είναι το μήνυμά μου σήμερα. Ευχαριστώ. Όντως, Προωθούμε αυτή την ιδέα ενίσχυση του συντονισμού ανάμεσα στις αρχές επιβολής του νόμου, γιατί και πάλι πρέπει να ενισχύσουμε τον συντονισμό και την εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στον Πολ Κλέμπερ Φαντεμπράκ, που είναι υπεύθυνο για την ε, υγεία στο Business Europe. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Business Europe ε, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της που μας ε, καλέσατε να έρθουμε εδώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε και η κυρία Ζαλντεμόζε. Όντως, το θέμα της ασφάλειας δεν είναι προαιρετικό, είναι υποχρεωτικό. από τον νόμο πρώτα απ' όλα. Και είναι και μια λογική ευθύνη που έχουμε απέναντι στους πολίτες μας. Όμως είναι καλό και για τις επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις για να επιβιώνουν χρειάζονται καταναλωτές. Άρα οι περισσότερες επιχειρήσεις δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην εικόνα που έχει προς τα έξω η επιχείρησή τους, το σήμα Και δεν θέλουν να παίρνουν, να αναβάνουν κινδύνους όσον αφορά την ε, ευθύνη που έχουν απέναντι στα προϊόντα. Αναγνωρίζουν λοιπόν και επιχειρήσει ότι η ασφάλεια είναι must, είναι υποχρεωτικό. Αλλά πρέπει να υπάρχουν μέτρα που να βοηθούν και τι επιχειρήσεις. Αναλογικότητα δηλαδή, νομική ασφάλεια, ευελιξία. Όσον αφορά την αναλογικότητα πρώτα απ' όλα. Εδώ δεν πρόκειται μόνο για τις δικαστικές ε, πτυχές. Πρόκειται για το επίπεδο της ε, ασφάλειας. Βλέπετε μερικές φορές λένε οι άνθρωποι δεν μπορεί να υπάρξει κανένα συμβιβασμός». Εγώ δεν νομίζω όμως ότι είναι σωστό αυτό, γιατί στην πραγματικότητα ο καθένας από εμά βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βαθμό κινδύνου καθημερινά στην καθημερινή του ζωή. Κανείς ε, δεν θεωρεί, υποχρεωτι... δεν θεωρεί ότι θα έπρεπε να πηγαίνουμε 0 χιλιόμετρα την ώρα στο αυτοκίνητό του για να αποφύγει τον παραμικρό κίνδυνο. Εννοείται πως αυτό δεν το θέλει κανείς. Οπότε ναι ε, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, είναι must, αλλά είναι και θέμα πολιτικής επιλογής. Άρα λοιπόν οι πολιτικοί πρέπει να πάρουν την ε, σωστή απόφαση και να την κάνουν νόμο. Και αυτό θα γίνει βέβαια λαμβάνοντα υπόψη τις ε, αρχές των εθνικών αρχών, τις αρχές επιβολής, για να μάθουν και οι πολιτικοί μας εδώ πώς θα επιβληθεί η όποια απόφαση πάρουν. Έπειτα να υπολογίσουμε ε, το κόστος και το όφελος από κάθε μέτρο ασφάλειας. Για παράδειγμα, ε, μπορεί να περιοριστεί ο βαθμός επιλογής που έχουν οι καταναλωτές, μπορεί να αυξηθούν οι τιμές. Πρέπει να δούμε και την ε, η ισορροπία σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ανάλογα με το από πού προέρχεται κάθε επιχείρηση. Εντάξει, μείωση του κινδύνου. Ναι, αλλά ο κίνδυνο μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να είναι και μικρό. Πρώτα απ' όλα, ζημιά που μπορεί να γίνει, μπορεί να είναι ε, μεγάλη ή μικρή. Όλοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να μην ε, βρεθούν σε μεγάλο κίνδυνο, αλλά δεν ξέρω αν είναι όλοι διατεθειμένοι να πληρώσουν πολύ περισσότερα για ένα πολύ μικρό ποσοστό κινδύνου, το οποίο θα μπορούσε ο καταναλωτής από μόνος του να διαχειριστεί. Χρειαζόμαστε ομοιόμορφους κανόνες που ομοιόμορφα να εφαρμόζονται στην αγορά μας. Πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να κάνουν αυτό που έχει αποφασιστεί. Πράγμα το οποίο όμως δεν γίνεται πάντα. Άρα χρειάζεται μια καλή διαδικασία επιβολής. Κάτι άλλο και χαίρομαι που το είπε και η κυρία Σαλτεμόζε, είναι ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του GSPD. έχει να κάνει με τις διασυνοριακές αγορές. Σίγουρα χρειάζεται συνοχή και σαφήνεια. Τα αναρμονισμένα προϊόντα που ανταποκρίνονται σε όλες τις προδιαγραφές, υπάρχει και σχετική οδηγία, δεν πρέπει να υποβάλλονται σε επιπλέον απαιτήσει βάσει του GPST, εκτός εάν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος εφόσον διατεθεί το προϊόν στην αγορά. Και τέλο έχουμε ήδη πει πολλές φορές μέχρι τώρα και χαιρόμαστε να το ακούμε, όλοι συμφωνούμε, ότι η επιβολή είναι ζωτική σημασία, γιατί τότε υπάρχει δικαιοσύνη απέναντι σε όλους μας. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία δεν έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θέλουμε. Γιατί αν αφήσουμε τους ε, ασυνείδητους εμπόρους να κάνουν ό,τι θέλουν, τότε αυτό είναι χειρότερο για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο Γιάνντε Κόνινγκ έχει τώρα το λόγο που είναι πρόεδρος του Φόρουμ Επιβολής του ΠΟΣΕΙΦ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και ε, του θέματος, αλλά αυτή δεν είναι η αρχή, η πρώτη μου διαφάνεια. Όπως βλέπετε έφερα διαφάνειες για να σας διασκεδάσω. Είμαι ένας από αυτούς τους officers που αναφέρατε εδώ και κάποιο καιρό ε, που καταρχήν η λιγότερο σημαντική διαφάνεια σας δείχνει ποιος είμαι. Αν θυμάστε μόνο από μένα πως ε, δουλεύω από το 96 ως ε, ε, υπεύθυνο για την εποπτεία της αγοράς, νομίζω αυτό θα αρκεί. Ε, στο Βέλγιο εννοώ. Εδώ αντιπροσωπεύω την ε, Base Safe που είναι μια οργάνωση που αποτελείται από όλους τους επόπτες της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Το 1990 δημιουργήθηκε αυτός ο οργανισμός και από το 2006 Ε, αποτελούμε την πλατφόρμα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια των καταναλωτών και την εποπτεία της αγοράς. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις επαφές μας και το συντονισμό μας για να βελτιώσουμε την ε, ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Η εποπτεία της αγοράς είναι σημαντική όχι μόνο για να έχουμε ασφαλή προϊόντα στην αγορά, που είναι ένας από τους τρεις τομείς που είναι σημαντικοί, αλλά επίσης, όπως ε, σίγουρα θα έλεγε και ο συνάδελφος δίπλα μου, για να δημιουργηθεί ισότιμο πεδίο για την ε, τις επιχειρήσεις και για να εξασφαλίσουμε την ε, ελεύθερη ροή των προϊόντων ασφάλεια το καταναλωτή είναι ένα δικαίωμα καταναλωτικό. Το να δημιουργηθεί ένα ισότιμο πεδίο και ασφαλή προϊόντα δίνει εμπιστοσύνη στον καταναλωτή, κάτι που σίγουρα ωφελεί την Ένωση και ε, οικοδομεί την εσωτερική αγορά. Ποιε είναι οι βασικές προκλήσεις λοιπόν για τις ε, αρχές εποπτείας αγορών. Καταρχήν να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε συνοχή ορισμοί, υποχρεώσεις, κίνδυνοι, έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να τα ερμηνεύει όλα αυτά με τον ίδιο τρόπο. Επίσης πρέπει να έχουμε κοινού πόρου ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν πολλούς ανθρώπινους πόρους, άλλοι έχουν εχουν υλικού πόρους, άλλοι έχουν οικονομικούς πόρους. Πάντοτε είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλου αυτού του πόρου και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Και επίσης πρέπει να φτιάξουμε ε, τις δυνατότητες για δοκιμές, ελέγχους, να δημιουργήσουμε τεχνογνωσία και καλύτερη πρακτική. Για να γίνουν όλα αυτά, Ε, με χαρά λάβαμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2006 και έπειτα. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ε, μεταμορφώσει την Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Έχουμε 19... 19 δράσεις για τα προϊόντα τα τελευταία πέντε χρόνια, κοινέ δράσεις ε, Πολλά κράτη-μέλη συμμετείχαν, συνήθως 20. Επίση, με χαρά μπορώ να σα πω ότι κάθε κράτο μέλο ε, συμμετείχε τουλάχιστον σε μία από αυτές τις ε, δράσεις. Όλοι λοιπόν ε, συμμετέχουν και αυτό που εντοπίσαμε κάνοντας αυτές τις κοινέ δράσεις είναι η ανάγκη για συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζουμε πως αυτό είναι ο, μόνο, μόνος λογικός και πρακτικός τρόπος για να εξασφαλίσουμε την καλή εποπτεία της αγοράς. Είμαστε ευτυχείς λοιπόν που τώρα πια υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για την εποπτεία ε, της αγοράς και φυσικά έχουμε συνδέσεις με τα τελωνία και επαφές με την Κίνα. Τώρα αυτή η διαφάνεια εδώ δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει πολλά ε, και γι' αυτό και έχουμε εδώ μικρά γράμματα για να χωρέσουν στη σελίδα. Αυτές είναι οι δραστηριότητες, να σας αναφέρω τις πιο πρόσφατες, ε, ας πούμε ε, τα προϊόντα τα οποία καλούν τα παιδιά, προκαλούν μάλλον τα παιδιά γιατί μοιάζουν με τρόφιμα, ε, τα solarium ε, και φυσικά πάντοτε έχουμε δράσεις για τα παιχνίδια. Ποια είναι τώρα τα διδάγματα που αποκομίσαμε από την εποπτεία της αγοράς. Καταρχήν η εποπτεία της αγοράς απαιτείται, όπως ακούσατε ήδη σήμερα, και από τη βιομηχανία και από τους καταναλωτές. Και γι' αυτό η συγκέντρωση των ανθρωπίνων και των υλικών πόρων ε, δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για την εποπτεία της αγοράς. Η συνεργασία, αν έχουμε το είδος συνεργασίας που χρειαζόμαστε, ευθυγραμμίζει την ερμηνεία των νομοθεσιών και την επιβολή αυτών. Πώς κάνουμε δηλαδή την εποπτεία της αγοράς, ποιες είναι οι κυρώσεις, πώς συνεργούμε... Αποτελεσματική λοιπόν εποπτεία της αγοράς κατά τη γνώμη μου είναι η συντονισμένη εποπτεία της αγοράς. Οι ανάγκες τώρα ε, θα ήθελα να πω τα εξή βασικά. Πρώτον, πρέπει να έχουμε κοινά στάνταρ, κοινέ προδιαγραφές για την εποπτεία της αγοράς. Ποιε είναι οι κυρώσει, οι διαδικασίε, η συχνότητα των επιθεωρήσεων. στη Γαλλία, α πούμε, λέει ότι ε, κάθε κατασκευαστή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά τα τρία χρόνια. Ε, αυτό θα πρέπει να το δούμε βέβαια σε συνδυασμό με τους πόρους που έχουμε και χρειαζόμαστε και μία νομική βάση για το συντονισμένη αυτή ε, εποπτεία επιθεώρηση των αγορών. Χρειάζεται λοιπόν οικονομική βάση και μακροπρόθεσμη δέσμευση. Έτσι νομίζω πως θα καταλήγαμε σε ένα οικονομικό, στηριζ, οικονομικός στηριζόμενο σώμα για την εποπτεία της αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ και να θυμίσω ότι πολλές από τις κοινέ δράσεις στο τέλος κατέληξαν σε κάποιο είδος ε, λήψης κοινών μέτρων, κοινοτικών μέτρων, όπως ας πούμε για τους αναπτύρες ή για την ε, υιοθέτηση συγκεκριμένων προδιαγραφών. Τώρα, έχω έναν κατάλογο μιλητών, αλλά πρέπει να σας δώσω ένα λεπτό στον καθέναν. Για διαφορετικά θα ξεφύγουμε από το χρόνο μας. Πρώτος είναι ο κύριος Τρολκίνσκι. Ιδέα. Yes. Go ahead. Today. Okay. Thank you. Sorry. Um, σας ευχαριστώ. Είναι μια ερώτηση περισσότερο για τη συντονίστρια. Αναφερθήκατε στα τρόφιμα στην εισαγωγή σας. Αναρωτιέμαι, μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ τα τρόφιμα, πώς μπαίνουν μέσα σε όλη αυτή τη συνολική στρατηγική και τι δράσεις προβλέπονται για τα διατροφικά συστατικά των τροφίμων. Συντονίστρια, προτείνω να ακούσουμε όλου του μιλητέ και μετά θα απαντήσουμε. Ο κύριος Τζορντάνο τώρα έχει το λόγο. Ε, ε, δεν είναι εδώ, λέει κάποιο άλλο από το κοινό, θα είναι όμω εδώ αργότερα. Ωραία. Η κυρία Τάουσα τώρα. Ευχαριστώ. Και εγώ μετά, αργότερα θα παρέμβω. Η κυρία Κρίς Τζοβάνι τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ότι εκτίμησα πολύ το γεγονός ότι τονίστηκε η επιβολή και ο συντονισμός. Πράγμα το οποίο τόνισε η Γενική Διευθύντρια Τεστόρη Κότζη. Φυσικά όλα αυτά σημαίνουν ε, και συντονισμό με όσους βρίσκονται επί τόπου, δηλαδή τις οργανώσεις των καταναλωτών, τις ενώσεις των καταναλωτών. Και θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα και κάποιες, ε, κάποια νούμερα. Εδώ και 40 χρόνια η Άλτο Κονσούμο συγκρίνει διάφορα προϊόντα και μεταξύ διαφόρων παραμέτρων έχουμε και την ασφάλεια. Το τελευταίο χρόνο, ανάμεσα στα διάφορα που έχουμε ε, ελέγξει, έχουμε ελέγξει έξι προϊόντα τα οποία είναι τουλάχιστον επικίνδυνα. Δηλαδή από κράνη σε αποσμητικά, ε, καθαρισμός ε, του νερού και μικρές ε, συσκευές, οικιακές συσκευές. Αλλά σχεδόν ποτέ στα 40 χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά δεν καταφέραμε να πετύχουμε την απόσυρση από την αγορά αυτών των επικίνδυνων προϊόντων. Το ερώτημα είναι λοιπόν γιατί. Ένα παράδειγμα θετικό ωστόσο, από τότε που άρχισε να ισχύει στη χώρα μας η οδηγία για τις ε, ε λανθασμένες πρακτικές, δηλαδή από το 2007 και μετά, καταφέραμε να κάνουμε 130 υποδείξεις στις αρχές εποπτείας ε, και παρενέβη στις μισές περίπου περιπτώσεις. Και εκεί έχουμε ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να διορθώσουμε τη στρέβλωση της αγοράς. Όμως, για να έρθω σε μια τρίτη πτυχή που αναφέρθηκε, νομίζω από τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προηγουμένως, Πιστεύουμε πως η Κομισιόν μπορεί να κάνει περισσότερα, να ασκήσει πίεση στα κράτη για να εγγυηθούν καλύτερη επιβολή. Όχι μόνο επιβολή, περισσότερη, αλλά καλύτερη, σωστότερη. Γιατί οι κυρώσεις όπως αυτές που συνδύεσαι η ε, ε, ε, αρχή εποπτείας με την ΕΠΟΛ για την νομοθεσία εγγύησης περί δεν είναι πρόβλημα μόνο ιταλικό αλλά ευρωπαϊκό κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Τζούελ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα παρακαλώ να πάρω το λόγο αργότερα. Η κυρία Μάρτιν Ρέι. Σας ευχαριστώ και θα είμαι σύντομη. Εδώ είμαι. Πολλά από τα θέματα ε, καλύπτονται στην πρότασή σας για την εποπτεία, για την ε, νομική αρρωγή, αντιπροσώπευση κτλ. Ακόμα και η συλλογική προσφυγή και η ενίσχυση του καταναλωτή είναι πράγματα που υπάρχουν και στη χώρα μου. Πολλές οργανώσεις στην Ευρώπη όμως ε, αγωνίζονται να επιβιώσουν. Ιδίως στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση που προκάλεσε το δημοσιονομικό σύστημα. Αγωνίζονται έτσι κι αλλιώς στις χώρες αυτές να μπορέσει ο καταναλωτής να έχει χρήματα να καταναλώσει και προσπαθούμε να πάρουμε και κάποια διδάγματα. Αγωνιζόμαστε σε καθημερινή βάση. Ο προπολογισμό έτσι κι αλλιώς, για τον καταναλωτή είναι μικρός. Πώς λοιπόν μπορούμε εμείς να αποφύγουμε ε, την εξαφάνιση κάποιων ε, οργανώσεων του καταναλωτή και πώς μπορούμε να δώσουμε νέα πνοή στον προπολογισμό για τις οργανώσεις αυτές που πλήττει τα ληστεία. Συντονίστρια. Δεν ξέρω αν είναι εδώ η κυρία Κιλελέκη που έχει ζητήσει το λόγο είναι για αυτήν τη στιγμή. Ε, θα ήθελα ε, πρώτα απ' όλα μία διευκρίνηση από την Business Europe ε, στο σημείο που αναφέρουν «Consumer safety is a must. Uh, business wants product to be safe customer expectations and responsibility to citizens. I would like some clarification. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. To citizens. Uh, το δεύτερο είναι, θα ήθελα να ρωτήσω την uh, Επιτροπή, ε, μέσα στην αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων είχαμε ζητήσει να υπάρχει ένα χωριστό κεφάλαιο το οποίο θα αναφέρεται στα σχολικά προϊόντα που, τον τελευταίο, που τα τελευταία χρόνια είναι κυρίως παιχνίδια. Θα ενταχθούν τελικά τα σχολικά προϊόντα με προδιαγραφές παιχνιδιών στην αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Και μία τρίτη ε, ερώτηση. Ε, όταν μιλάμε για κυρώσεις, για παραβίαση της ασφάλειας των καταναλωτών, ε, μιλάμε συνήθως για proportionality. Ε, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε ε, ότι αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτρεπτικές διότι κάποια στιγμή δεν, ε, κάποιες ζημίες δεν, έχουν, δεν μπορούν να αποζημιωθούν και θα σας φέρω ένα παράδειγμα θάνατο από μία ασφαλές ηλεκτρικό σίδερο από ηλεκτροπληξία αυτή, αυτή η ζημία δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει αποζημίωση. Άρα μήπως πρέπει να γίνουν πολύ πιο αυστηρές οι κυρώσεις ώστε να δρουν προληπτικά. Ευχαριστώ. Okay, Σας ευχαριστούμε. Καλώς. Υπάρχει κάποιος ευρωβουλευτής μήπως που θέλει να παρέμβει σε αυτό το στάδιο. Όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε ας ξεκινήσω να απαντήσω εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Την κυρία Χωσίνσκη πρώτα απ' όλα. Πώς ε, το Eurofood περιλαμβάνεται στην ατζέντα για τον καταναλωτή. Μα θέλουμε να καλύψουμε το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών που επηρεάζουν την καθημερινότητα των καταναλωτών. Γι' αυτό και συμπεριλαμβάνουμε και τις πολιτικές μας για τα τρόφιμα, γιατί θέλουμε ο καταναλωτής να αντιληφθεί τι δουλειά γίνεται στον τομέα των τροφίμων. Βέβαια, η εκπόνηση των κανόνων μας πιστεύω ότι είναι καλή. Ρωτήσατε κάτι και με για τα συστατικά τροφίμων. Έπειτα να ρωτήσω την κυρία Τζοβάνη. Αναφερθήκατε σε περιπτώσεις όπου βρέθηκαν κάποια ψηλά ε, ποσοστά σε ορισμένα προϊόντα. Εδώ είναι οι εθνικές αρχές οι οποίες πρέπει να ξεκινήσουν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Οπότε φαντάζομαι ότι οι δικές σας αρχές εξετάζουν την υπόθεση και αν δεν έκαναν τίποτα είναι γιατί δεν θεώρησαν ότι υπήρχε κίνδυνος. Όσον αφορά τώρα τη στήριξη των οργανώσεων καταναλωτών. Ναι, συμφωνούμε ότι υπάρχει πρόβλημα σήμερα που είμαστε στην οικονομική κρίση, πώς θα συνεχίσει να είναι ισχυρή η φωνή των καταναλωτών. Εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις οργανώσεις των καταναλωτών και μέσα στο νέο πρόγραμμα θα αυξήσουμε τη στήριξη στις οργανώσεις καταναλωτών και μπορούμε να κάνουμε έκκληση έτσι ώστε οι οργανώσεις ε, των καταναλωτών να στηριχθούν και σε εθνικό επίπεδο. Γιατί εμεί χρηματοδοτούμε ό,τι έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, για την κυρία Κιλελέκη, για το κατά πόσο θα υπάρξει η ειδική κάλυψη και των προϊόντων που κυκλοφορούν στα σχολεία, η προσέγγιση μας είναι ότι πρόκειται για μια οριζόντια οδηγία και υπάρχουν ειδικέ οδηγίες για κατηγορίες, για τα παιχνίδια για παράδειγμα και θα δούμε κατά πόσο πρέπει να υπάρξει και κάποια ειδική οδηγία για τα προϊόντα αυτά τα σχολικά. Υποβλήθηκαν ερωτήσεις και σε άλλους ομιλητές, οπότε το ProSafe ή EuroBusiness Business, παρακαλώ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ερώτημα το τι σημαίνει ευθύνη των πολιτών. Σας έδωσα τους ε, λόγους της, ε, των επιχειρήσεων γιατί πρέπει τα προϊόντα να είναι ασφαλή. Δεν θα το επαναλάβω. Όταν αναφέρομαι στην ευθύνη των πολιτών τώρα, είμαστε ευτυχώς σε μια κοινωνία όπου δεν είναι όλοι κάποια στιγμή ληστές όταν είναι υπεύθυνοι για κάποια εταιρεία. Ε, καταλαβαίνω λοιπόν ότι αν τα προϊόντα τους δεν είναι ασφαλή, η υπηρεσία τους δεν είναι ασφαλή, έχει αυτό επιπτώσεις για τους άλλους συμπολίτες τους. Ε, δεν γίνεται αυτό πάντα και παντού. Είναι κάτι που εξαρτάται και από τον ε, τις παραδόσεις μιας χώρας και γι' αυτό είναι σημαντικό η ε, δημοσκοπήσεις των αγορών και όχι μόνο δημοσκοπήσεις αλλά και συντονισμένες δημοσκοπήσεις γιατί οι, οι, οι αλυσίδες ε, προμήθειας ε, και αγοράς έτσι κι είναι διεθνή σήμερα. Ήμουν σε μια ομάδα γιατί κάνω κάποια σεμινάρια για την ε, ηθική επιχειρήσεων αν θέλετε που γίνεται κάθε χρόνο και έτσι μπορούμε να προωθήσουμε την ευθύνη προς τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Μία σύνομη απάντηση. Αυτό που αναφέρθηκε για τι δημοσκοπήσει των αγωνών και τι οργανώσει των καταναλωτών. Θέλω να πω ρητά ότι δεν ακούμε μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τις οργανώσεις των καταναλωτών και είμαστε πάντα πολύ ευτυχεί αν μας δίνουν πληροφορίε για κάποια προϊόντα που ίσως δεν είναι ασφαλή. Όπω αναφέρθηκε, το σύστημα που ακολουθούμε λαμβάνει υπόψη. Δηλαδή ότι εάν ληφθούν μέτρα για μία χώρα θα ληφθούν μέτρα για όλες τις χώρες. Και τώρα για τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αναλογικές αλλά και αποτρεπτικές. Αυτό σημαίνει δεν γίνεται πάντα η ανάκληση των προϊόντων, αλλά έχουμε και άλλα μέτρα. από σειρή, παραδείγματο χάρη, διακοπή της παραγωγής, πληροφορίες προς τους καταναλωτές κλπ δεν είναι πάντα δράση υψηλή ορατότητα, δηλαδή το επειδή δεν το είδατε δεν σημαίνει ότι δεν έγινε τίποτα. Ευχαριστώ κύριε Νόλ. θέλετε να μιλήσετε. Ε, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πια πεπισμένη ότι πολλά μπορούν να γίνουν για να βελτιώσουμε το σύστημα ε, νομοθεσία, εντονισμός, ε, διάλογος κλπ. Θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε γρήγορα. Ευχαριστώ. Πρώτος ευχαριστώ. Δύο λόγια, για να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια του καταναλωτή, χρειαζόμαστε κανόνες και επιβολή των κανόνων επίσης. Μάλκο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάολα. Περνάμε τώρα στην, ε, στο επόμενο σημείο και καλώ στην πλατφόρμα. σου πρέπει να είσαι από την That is our disabled lift button. so, um, so I'm really pleased to welcome our second Director General from the Commission. We have a, great team with us today in this joint hearing. Καλώς ήρθατε λοιπόν δεύτερη γενική διευθύντρια εδώ για δικαιώματα, βασικά δικαιώματα, για δικαιοσύνη βασικά δικαιώματα και τους πολίτες. Καλώς ορίζω εδώ Όποιος θέλει να μιλήσει τώρα ή μετά από τους συμμετέχοντες, στείλτε μας ένα σημείωμα ή το επισκεπτήριό σας για το ποιος είσαι, ποιον εκπροσωπείτε και πού θέλετε να μιλήσετε. Ο Τζιάννο και η Μπιάνκα εδώ πέρα μαζεύουν κατάλογο με όλους τους ενδιαφέρον να μιλήσουν. Βέβαια οι ευρωβουλευτές καλούνται ούτως ή άλλως να συμμετάσχουν. Θα Θέλουμε βέβαια κατά το πολύ να συμμετάσχουν. Φιλοσφά, θα σου δώσω το λόγο τώρα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Μάρκο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαι εδώ και μπορούμε να συζητήσουμε ειδικέ πτυχέ ε, τη ατζέντα για τον καταναλωτή, νομοθεσία δηλαδή. όχι μόνο την ε, νομοθεσία αλλά και την επιβολή της ε, νομοθεσίας αυτής. Η νομοθεσία πρέπει να υπάρχει γιατί ε, αλλάζει το, το περιβάλλον της κατάλληλος. Παραδείγματος η ψηφιακή περίοδος στην οποία ζούμε συμβάλλει διαφορετικά. Επίσης και για τους καταναλωτές θα πρέπει να ροδοτορηθούμε κατά πόσον πρέπει να αλλάξει ε, γι' αυτό και η νομοθεσία για τους καταναλωτές. Και μετά βέβαια καλό είναι να έχουμε ισχυρή νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα επιβληθεί αυτή η νομοθεσία. Και από ό,τι κατάλαβα η αντιπρόεδρος κυρία Ρέντινγκ ανέφερε το θέμα σήμερα το πρωί, άλλωστε ήταν χρήσιμο να το συζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Έχουμε θαυμάσιο πάνελ εδώ ε, ατόμων που εκπροσωπούν διάφορε αρμοδιότητε. τον Τόμα Νότφρετ από την, ε, το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών και που θα μας πει ποιε σκέψεις υπάρχουν στη χώρα του όσον αφορά την νομοθεσία για τον καταναλωτή ιδίω σε ένα ψυχιακό κόσμο. Έχουμε τον Τζίζεν Φρήμαν που είναι από την ΟΕΦΤΗ και συμπληρώνει τα διάφορα αυτά σημεία για τις αθέμητες πρακτικές. Έχουμε τη Μαρία Ρηγογέν Περές, Ευρωβουλευτή, που είναι η συγκήτρια για τους ευάλωτους καταναλωτές και αυτή είναι μια οπτική στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Και μετά έχουμε τον Ροντρίγιο Γκουβέια. που θα αναφερθεί στο θέμα τη αϊφόρου κατανάλωση και που εκπροσωπεί εδώ ως Γενικός Γραμματέας την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιρισμών Καταναλωτών. Και μετά έχουμε τον Ανδρέα Σβάπ, που είναι εδώ, ναι, που θα είναι και ο πρώτος ομιλητής στο πάνελ αυτό και θα αναφερθεί στο, στο θέμα της νομοθεσίας της πωλήσει μια πρωτοβουλία της Κομισιόν και ιδίως όσον αφορά τις πτυχές που αφορούν τον καταναλωτή. Παρακαλώ, κύριο Σφάβ, έχει το λόγο. Αγαπητοί Φρανσουάς, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και τις νομικές πτυχές της νομοθεσίας για τους καταναλωτέ. Ήδη κάποια ακούστηκαν για το θέμα αυτό και γι' αυτό εξ τη ομάδα του ΕΛΚ θα ήθελα να αναφερθώ σε τρει βασικέ αρχέ που κατά τη γνώμη μα είναι αποφασιστικότητα για την περαιτέρω εξέλιξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην Ευρώπη. Καταρχήν, θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο απόλυτα διαφανεί κανόνε. Δεύτερον, η εφαρμογή στην ε, εκάστοτε εθνική νομοθεσία να ελέγχεται προσεκτικά και να φροντίσουμε αυτό το δίκαιο που έχει αποφασιστεί να εφαρμόζεται και σωστά. Ε, στις γρήγορη συμβουλή μου θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στην ίδια την οδηγία για τους καταναλωτές. Η κυρία Ρέντινγκ αναφέρθηκε προηγουμένως ότι από 18 τομείς που πρόκειται να εναμοστικούν πλήρω, έχουν ενωπηθεί 5 ως 7. Δηλαδή σε αυτούς τους τομείς έχουμε σαφείς κανόνες. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε ότι και η εφαρμογή στα κράτη-μέλη θα πρέπει να ελέγχεται εξίσου προσεκτικά και νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολείται με μία σειρά ε, άλλων προτάσεων δεν μπορεί να εξετάζει τόσο προσεκτικά το θέμα της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία όπως το έκανε στο πρώτο ήμιση της ε, θητείας. Το τρίτο θα πρέπει οι κανόνες που υπάρχουν να εφαρμόζονται και σωστά. Σε ένα δεύτερο βήμα η Κομισιόν προτείνει ένα 8ο καθεστώς, δηλαδή το λεγόμενο Consumer Contract Law, το, το για τις κατανοητικές συμβάσεις. Γιατί είδαμε ότι η συνοδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή στο παρελθόν με πολλά κράτη-μέλη δεν πετύχαμε ε, ομοιόμορφη μεταφορά και τώρα αυτή η ισοτιμία επιτυχάνεται γιατί τη χρειαζόμαστε για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Οι συζητήσεις είναι πως θα πρέπει να ε, εκτιμήσουμε την πρόταση αυτή για το 28ο καθεστώς. Ο συνάδελφος Σαν Πέτερ Μάγερ έχει ξεκινήσει την εργασία του, τίθενται όμως διάφορα ερωτήματα που αφορούν την συνοχή μεταξύ της οδηγίας για τους καταναλωτές και της πλήρωσης εκεί ε, εναρμονισμένες διατάξεις και τη νέα αυτή πρόταση. Δεν θα επιστάσει στις λεπτομέρειες, αλλά το Κοινοβουλίο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ότι η ε, νομοθεσία που έχει ήδη εγκριθεί να περάσει στην νέα αυτή νομοθεσία και να επικαλύπτει με αυτή. Ταυτόχρονα όμως να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω με το ε, ενιαίο δίκαιο για τους καταναλωτές και να δουν τα κράτη-μέλη αν θέλουν την αρμόνιση ή αν δεν τη θέλουν. Δεν μπορούν να λένε όχι σε όλες τις προτάσεις Κομισιόν βέβαια. Ταυτόχρονα θα ήθελα εδώ να αναφέρω θετικά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει πολλές δυνατότητες ευελιξίας να επιτρέψει δηλαδή να ακούσουμε τις απόψεις των κρατών μελών, δηλαδή στον οδικό χάρτη Αναφέρεται και ένας ενιαίος νόμος ενδεχομένω για τις πωλήσει εφόσον χρειάζεται κάτι τέτοιο. Όλοι λοιπόν που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν προτεραιότητές τους και όλοι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τοποθετηθούν. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τους ε, στηρίξει με κάθε δυνατότητα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ριγογέν Πέρες έχει τώρα το λόγο για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Φρανσουάς. Θα αρχίσω αναφερόμενοι σε αυτό το οποίο είπες, ότι οι καταναλωτές ε, αλλάζουν και θα αλλάζουν με τον ψηφιακό κόσμο. Και ο συνάδελφος ΣΒΑΠ είπε επίσης ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά όσον αφορά τα δικαιώματα. Το 1975 δημιουργήθηκε το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών Εκεί συμπεριλαμβανόταν ε, ένας κατάλογος πέντε βασικών δικαιωμάτων για τους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια από τότε έχει κάνει μεγάλο δρόμο και έχει ετοιμάσει ένα πλαίσιο προστασία των καταναλωτών. Όμως η νομοθεσία για την ανάπτυξη της ε, ενιαίας αγοράς προχώρησε πιο γρήγορα από ότι η προστασία των καταναλωτών. Συνεχίζουμε βέβαια να προχωράμε και να συμπεριλαμβάνουμε όλο και περισσότερα δικαιώματα των καταναλωτών για να ενισχύσουμε την ευημερία τους, κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην παρετέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για το 2020. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι καταναλωτές δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα, αλλά στα γενικότερα πλαίσια υπάρχει μια ε, κατηγορία πολύ ειδικοί μεταξύ των καταναλωτών, που είναι οι ευάλωτοι καταναλωτές. Ε, αυτοί λοιπόν απαιτούν ειδική αντιμετώπιση, ειδική προστασία και ειδική ε, αντιμετώπιση από πλευράς των αρχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και αντιλαμβάνεται ότι είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι καταναλωτές για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, εδωγενείς κλπ, ε, οι οποίοι μπορεί να πλήξουν οποιονδήποτε από εμά. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Μπορεί κάποιος να είναι ευάλωτος εξαιτία ενός παράγοντα ή πολλών. Το θέμα λοιπόν αυτό του ευάλωτου του καταναλωτή αναφέρεται στην οδηγία του 2005 για τις εμπορικές αθέμητες πρακτικές των επιχειρήσεων σε σχέση με τους καταναλωτές της εσωτερικής αγοράς. Αναφερόμενοι στο καθεστώς αυτό του ευάλωτου καταναλωτή, αναφέρονται διάφορες πρακτικές οι οποίε μπορούν να πλήξουν ένα καταναλωτή, ο οποίο δεν είναι αρκετά μημένο, αρκετά ενημερωμένο. Πρέπει να προστατεύσουμε και το οικονομικό όμως συμφέρον των καταναλωτών, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει και η υγεία του, υπάρχει η ηθική του αξιοπρέπεια κλπ. κλπ. Η οδηγία λοιπόν για την προστασία των καταναλωτών πάνω στην οποία δούλεψε ο συνάδελφος ΦΑΠ από την ΙΚΟ δεν εφαρμόζεται για ορισμένους τομείς όπου οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και ότι υπάρχει ειδική ρύθμιση σε μερικές περιπτώσεις. Απλώς στο σημείο 34 κάτι αναφέρεται. Όμως πρέπει να υπάρχει προσεβατική ενημέρωση αλλά και μετά. Και εφόσον ο προμηθευτής ή ο πολιτής δεν τηρεί τον νόμο να μπορεί να επιστρέψει εύκολα το προϊόν ο καταναλωτής. Στην πρόταση κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 μιλάει για τη βελτίωση της διαπαιδαγώγησης και της ενημέρωσης των καταναλωτών, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματά τους και οι τρόποι προσφυγής που έχουν για να τηρούνται τα δικαιώματά τους και διασυνοριακά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια φιλόδοξη πρόταση η οποία συμπεριλαμβάνει και την ε, κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα μιλάει για τους ηλικιωμένου. και λέει ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στην κοινωνία και να αποτελούν ε, αυτόνομους παράγοντες της αγοράς. Ναι, μεν ε, αναφέρονται αυτά, αλλά δεν επαρκούν, γιατί δεν καλύπτουν όλους τους ευάλωτες καταναλωτές. Εξάλλου στην πράξη, έχει φανεί ότι από μόνη της η ενημέρωση δεν φτάνει για να ενισχύσει τον καταναλωτή. Θα σταματήσω εδώ γιατί έχει περάσει ο χρόνος μου και μετά κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα παρέμβω και πάλι. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Νόβιτς τώρα έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να συνδυάσω και να, σε, να παρουσιάσει 3 λεπτά μια ομιλία δέκα λεπτών. Το θέμα είναι ότι ένας καταναλωτή δεν είναι μόνο καταναλωτή, είναι και ένας παίκτη αγοράς. Θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη όταν εξετάζει κανένας τον καταναλωτή. Δηλαδή ο καταναλωτή δεν είναι μόνο κάποιος που χρειάζεται προστασία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Επίση, ο καταναλωτή δεν είναι μόνο καταναλωτή όταν πάει μέσα στο, ε, ε, στο διαδίκτυο, αλλά είναι και χρήστης, είναι και πολίτης και Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το τι κάνουμε στην ε, Νορβηγία για το θέμα αυτό. Δεν είχαμε πολύ μεγάλα ε, προϊόντα με το Facebook, γιατί ο καταναλωτή δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να υπάρχει μια ομάδα Facebook κατά της ε, για την προσοχή του καταναλωτή περνώντας δηλαδή τώρα από τα αγαθά στην, στις υπηρεσίες, βλέπετε ότι κανένας αγοράζει κάτι και το βάζει μετά στο διαδίκτυο και αυτό αλλάζει ανάλογα με τις ενημερώσεις που του κάνει. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι διαπραγματεύσιμο για το καταναλωτή. Είχαμε στην Νορβηγία με υπόθεση με τη Sony, η οποία ε, προσέφυγε στον διαμεσολαβητή ότι κάποιοι ε, παρενέβησαν στο διαδίκτυο και κατέστρεψαν 3 εκατομμύρια PlayStation. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί κανάς να πατήσει ένα κουμπί και να αλλάξει τα πάντα μέσω σε αυτό που ε, χρησιμοποιεί ε, ο, ο, ο πολίτης. Μπορεί κανάς να αφαιρέσει τα περιεχόμενο από προσωπικά βίντεο πολλά και πολλά και άλλα. Και αυτό είναι κάτι που δεν έχει α, ακόμα, δηλαδή αυτός ο διτός μονόλογος, αν μπορώ να σας το πω, προς τις δύο κατευθύνσεις. Και γι' αυτό δεν, χρειά, δεν αρκεί ένα συμβατικός νόμος ή νόμος επί των συμβάσεων, αλλά χρειάζεται να υπάρχει διακανονισμή. Γιατί αλλιώ, ε, αν υπάρχουν νομικοί ε, κανονισμοί, θα καταστρέψει παραδείγματο τον με ό,τι κάνει. Επίση, ο καταναλωτή ε, χρειάζεται δυνατότητα στην αγορά. Ο διακανονισμό όπου υπάρχει πνευματικά δικαιώματα, νομοθεσία για τον ανταγωνισμό κλπ. Όλα αυτά είναι τμήμα της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Το θέμα της εμπιστοσύνης αναφέρθηκε πολλές πολλές φορές. Αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι κάτι καινούριο. 20 χρόνια είχαν μπροστά τους οι επιχειρήσεις και έδειξαν ότι μπορούν πραγματικά να συμπεριφερθούν σωστά και ακόμα συζητάμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Αν δεν κάνουμε τίποτα υπάρχουν τεράστιες απώλειες. 46 δις, αν δεν κάνω λάθος, α, χάνονται. αυτά είναι τα στοιχεία που δίνει το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, το Τμήμα Οικονομολογίας από πέρσι. Και αυτό έχει, όπως είπαμε, και ουσιαστικές ε, και νομικές ε, ε, επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστούμε. Πράγματι σε τρία λεπτά προσπάθησα να τα πεις όλα. Ο κύριος Φρέιμαν έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες ε, διαφάνειες οι οποίες ίσως θα βοηθήσουν. Είμαι λοιπόν νομικός διευθυντής ε, στο OFT και ασχολούμαι με το νοχικό δίκαιο. Ένα από τα πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε πρόσφατα είναι ε, η νομοθεσία για τους καταναλωτές, γιατί υπάρχει και κατά πόσο αυτό βοηθάει τις αγορές. Τι εννοούμε. Δεν εννοούμε μόνο την προστασία των καταναλωτών, εννοούμε και προστασία της οικονομίας, έτσι ώστε η οικονομία να λειτουργεί αποτελεσματικά. Και θέλουμε οι ευρωπαϊκές και οι βρετανικές επιχειρήσεις να λειτουργούν αποτελεσματικά. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι πρέπει το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο για όλου, για την κοινωνία συνολικά. Και είναι πολύ σημαντικό όταν σκεφτόμαστε την αξιολόγηση. Δηλαδή την κάθε περίπτωση που εξετάζουμε έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Συχνά η προστασία των καταναλωτών έχει να κάνει με, τους, ε, με τις απάτες που γίνονται πολλέ φορέ από του εμπόρου, την αναποτελεσματικότητα, στη διανομή, στην παραγωγή, στην πώληση. Και αυτό γιατί έχει να κάνει με όλου, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μα. Και όντω, εξοργιζόμαστε με αυτό. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε τις αγορές μας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Ποιο είναι το οικονομικό πλαίσιο τώρα, αυτό μας ενδιαφέρει. Θέλουμε αποτελεσματικότητα στην αγορά. Έχουμε κάνει κάποιες μελέτες όπου μελετούσαμε τις συμβάσεις και τις διαφημίσεις προϊόντων, συμβάσεις με τους καταναλωτές δηλαδή και διαφημίσεις προϊόντων. Και σκεφτόμαστε και τι επανόρθωση μπορούμε να έχουμε. Δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι τέλειο, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι καταναλωτές μπορούν πάρα πολύ ε, λογική, για παράδειγμα όσον αφορά την επανόρθωση, μερικές φορές ο καταναλωτής αν είναι να χάσει 15 λίρες δεν θα κάτσει να μπει στη διαδικασία της προσφυγής για να πάρει πίσω τα λεφτά του. Έπειτα καμιά φορά δεν έχει διαβάσει το συμβόλαιο καλά ο καταναλωτής και αυτό το λένε οι δικαστές. Αν δεν έχει διαβάσει το συμβόλαιο ε, δεν μπορείς και να δικαιωθεί. Ναι, αλλά όταν κάποιο περιμένει σε ένα μαγαζί να ψωνίσει και του λένε ότι πρέπει να διαβάσει τον κανονισμό και έχει ολόκληρη ουρά από πίσω, τι θα κάνει, πόσο χρόνο θέλει για να κάτσει να το διαβάσει αυτό. Ε, δεν πρέπει να τιμωρείται επειδή δεν έχει διαβάσει όλο αυτό τον κανονισμό. Δεν θέλουμε λοιπόν να κατηγορούνται γι' αυτό οι καταναλωτέ και να τιμωρούνται γι' αυτό. Πρέπει να δούμε επίση και το κοινωνικό κόστο. Δεν θέλουμε να υπάρχει μια διαστραβόμενη. Ε, επιδότηση κατά κάποιο τρόπο της αγοράς. Πολλές φορές είναι σαν ε, ε, δέλτα αυτούς οι οποίοι πληρώνουν σε ένα γυμναστήριο και τελικά δεν πηγαίνουν και χάνουν τα λεφτά τους. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που σκεφτόμαστε είναι τελικά ο νόμος έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε και ως δικηγόροι, ως νομικοί αυτό ακριβώς προσπαθούμε να δούμε. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι δραστήριος γιατί ο καταναλωτής δεν είναι μόνο κάποιος ο οποίος πηγαίνει και αγοράζει ένα παντελόνι μια μπλούζα, είναι και κάποιος ο οποίος ανάλογα με τις αγορές του εκείνη και τα νήματα της αγοράς. Στο eBay δείτε τι γίνεται. Άρα λοιπόν είναι ένας καταναλωτής οικονομικά δραστηριο. Ε, ο οικονομικά δραστηριο Καταναλωτή δεν προστατεύεται αρκετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε λιγάκι τον ορισμό που χρησιμοποιεί το UCPD στις διάφορες περιπτώσεις και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι απεφάνθη στην περίπτωση Casa Dental Kit. Δεν είναι λογικά αυτά αν λάβουμε υπόψη μας ε, τον καταναλωτή ο οποίος είναι οικονομικά δραστήριος και πουλάει είτε ένα αυτοκίνητο είτε κάτι άλλο, δεν είναι... Ίσως θα έπρεπε ο καταναλωτής να μην περάσει από μια κατάρτιση για να γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά του. Και αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε, να έχει ο καταναλωτής ε, νέες ευκαιρίες. Εδώ είναι που ο νομοθέτης πρέπει να ξεκοιτάξει τον ορισμό του καταναλωτή για να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου αυτοί οι οποίοι είναι οικονομικά δραστήριοι τελικά χάνουν από την αγορά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και συγγνώμη που τα είπα τόσο γρήγορα, λέει ο μιλητής. Thank Good morning, Είμαι ε, είμαι από την ε, Eurocop που εκπροσωπεί μια σειρά συνεταιρισμών ε, των καταναλωτών. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θα σα μιλήσω για την εφορία. Τι σημαίνει εφορία, τι θέλει ο καταναλωτή. Αυτό που θέλει είναι η τιμή να είναι σωστή. Αλλά τιμή χαμηλή τηρώντα κάποια πρότυπα. Ασφάλεια ποιότητα και αηφορία. Όχι μόνο όσον αφορά το περιβάλλον, αλλά και κοινωνικά παραδείγματο χάρη. Για επιταυτεί αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν το κατανοητή για τα επόμενα έτη να εξετάσει το, το θέμα της αηφόρου κατανάλωσης και παραγωγής η Κομισιόν προετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης για το τομέα αυτό και θα μπορούσε εδώ να είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ανησυχίες των καταναλωτών να ενσωματωθούν σε αυτές τις πολιτικές της αηφορίας. Γιατί παρόλο την οικονομική κρίση, παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, η αηφορία δεν μπορεί να παραβλεφθεί. ούτως αναφορά αφορά το τομέα του περιβάλλοντος, γιατί οι καταστροφές που φέρουμε στο περιβάλλον δεν μπορούν εύκολα να ε, καλυφθούν και επίσης και η κοινωνική αηφορία είναι ένα σημαντικό θέμα. Βλέπουμε καθημερινά οι καταναλωτές να επιθυμούν στα προϊόντα που αγοράζουν να τηρούνται οι αρχές της αηφορίας και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κριτήριο να λαμβάνεται εξίσου υπόψη όπως το κριτήριο της ασφάλειας. Γιατί για την ασφάλεια, όπως είπε προηγουμένως η Γενική Διευθύντρια είμαστε πάρα πολύ προχωρημένοι. Στην Ευρώπη, παραδείγματο χάρη, είμαστε στου καλύτερου στον κόσμο όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και υπάρχουν αυστηρά κριτήρια και έλεγχη. Όσον αφορά την αηφορία, δεν νομίζω ότι έχει επιδοθεί τόση πολύ μεγάλη σημασία και θα έπρεπε γιατί δεν είναι δίκαιο ούτε προς επιχειρήσεις ούτε προς τους καταναλωτές να πηγαίνει κάποιο εκτό Ευρώπη να παράγει τα προϊόντα του χωρί να σέβεται τα ίδια περιβαλλοντικά κριτήρια ή κοινωνικά κριτήρια, να έχει δηλαδή ένα αθέμητο οικονομικό πλεονέκτημα και μετά να πολλαλεί αυτά τα προϊόντα στις ίδιες αγορές όπως εκείνα που έχουν παραχθεί τηρώντας όλους τους αυστηρούς κανόνες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ χρόνο να τοθούν οι ανησυχίε των καταναλωτών στι άλλε πολιτικέ και βέβαια και η επιβολή των διατάξεων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα τη ε, συλλογική προσφυγή. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, δεν θα έχουμε ποτέ την σωστή επιβολή των νησιών των νόμων. Αλλά αυτό βέβαια θα μπορεί να γίνει εάν η αϊφόρος ανάπτυξη επανέλθει στα χέρια του καταναλωτή. Γιατί οι κατανόητε αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν να, πού έχουν πλεονεκτήματα από την οικονομική εξέλιξη. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα πλεονεκτήματα, τα ωφέλη από την αηφορία να έρχονται πίσω στα χέρια του καταναλωτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σα ευχαριστώ. Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Είχαμε πολλέ ενδιαφέρουσε παρουσιάσει. Ακούσαμε ότι υπάρχει ανάγκη για διαφανείς ε, κανόνες, για αυστηρή επιβολή, το θέμα των συλλογικών ε, προσφυγών. Ακούσαμε επίση ενδιαφέρουσε ιδέε όπω χάρη εξέταση των ορισμών ε, των καταναλωτών. Ακούσαμε διάφορα επίση προτεσία των καταναλωτών από τη σκοπιά των οικονομικών ενδιαφερόντων και ούτω καθεξής. Έχω ένα μακρύ κατάλογο εδώ ατόμων που θέλουν να παρέμβουν στα θέματα αυτά. Θα δίδωσω το λόγο σε όσους μπορώ για ένα λεπτό ο καθένας. Λοιπόν, ερώτηση. όχι δηλώσεις και ε, ομιλίες. Η κυρία Τός έχει το λόγο από το ECCG Germany. Tausch ist mein Nachname. Ναι, Τάος λέγαμε μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο σημείο. Ψηφιακός κόσμος. Αυτό σημαίνει επίσης ψηφιακό εμπόριο και είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ η προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Εγάζεται πάνω σε αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπάρχουν πάρα πολλά σχετικά στην ε, ατζέντα για τον καταναλωτή. Αυτό είναι λυπηρό, ανησυχητικό. Θα πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό να συμπεριληφθούν περισσότερα. Επίσης, αναφέρθηκε το ότι η νομοθεσία και η εφαρμογή και η μεταφορά της νομοθεσίας αυτής στο εθνικό δίκαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνο που παραβλέπετε είναι η εφαρμογή αυτών στην πραγματικότητα. Ιδίω πώς μπορεί για την προστασία των δεδομένων να υπάρχει ενημερωμένη συνένεση, πώς μπορούν να δοθούν όλες οι ενημερώσεις για τη συμβάση. Αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε στι επιχειρήσεις. Στην ε, τομέα της ε, προστασίας των δεδομένων υπάρχει το θέμα της ε, αυτοποχρέωση. Εδώ δεν εντάσσονται όμω ούτε οι ενό των καταναλωτών ούτε οι επιστήμονες και θα πρέπει να προωθήσουμε οι κανόνες που ε, υιοθετούνται να είναι στην πραγματική του εφαρμογή προς όφελο των καταναλωτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Um, a thread that's run through almost all Ευχαριστώ. Κάτι το οποίο διέπει όλε τι παρουσιάσει και τα σχόλια σήμερα το πριν είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη και ο ευάλωτο χαρακτήρα των καταναλωτών. Και πιστεύω επίση πω η πραγματικότητα είναι ότι αναμφίβολα η οικονομική κρίση ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για όλα αυτά. Γι' αυτό η δική μου παρατήρηση είναι ότι σε σχέση με τη στρατηγική για τους καταναλωτές, ε, εφόσον θέλουμε να προχωρήσουμε, μήπως θα ήταν πιο λογικό και ρεαλιστικό να χρησιμοποιήσουμε την πρόταση της κυρίας Έλτερ Μόζε που έγινε προηγουμένως ότι θα πρέπει δηλαδή κατά κάποιο βαθμό να βοηθήσουμε την ε, εφαρμογή και την επιβολή του νόμου που είναι αργή και δαπανηρή. Μήπως αυτό μπορούμε να το, να το διευκολύνουμε. Ιδιαίτερα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όπου χρειάζεται πρόοδος. Να γίνει μια συντονισμένη προσέγγιση προς το naming and shaming. Δηλαδή το να ονοματίζουμε τους ε, ε, δράστες, τους απαταιώνες. Ε, τελευταία μου ερώτηση είναι Μήπως είναι λογικό λοιπόν ρεαλιστικά να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία ώστε να αναθέσουμε στους ίδιους της ενός των καταναλωτών να το κάνουν αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φέλλερ. Food and Drink Europe. Um, Food Drink Europe represents the uh, Η Food and Drink Europe αντιπροσωπεύει την ε, βιομηχανία τροφίμων και ποτών ε, στην ε, Ευρώπη, της Ευρώπης και θέλω να απευθυνθώ στην ε, Διευθύντρια Λεμπάγη γιατί νομίζω ότι δεν μιλάμε αρκετά για το γεγονός ότι ο τομέας μας αντιπροσωπεύει πάνω από 300 εταιρείε που είναι μικρομεσαίες και η νομοθεσία περιπολίσεων ε, αφορά και τις, ε, τους αθέμητες συμβάσεις μεταξύ εμπόρων εγώ έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Πώς θα γίνει η νομοθετική πρόταση που θα, διέψει, θα διέπει μάλλον ε, τις σχέσεις ανάμεσα στις ε, εταιρείε. Ε, το 99% των εταιριών μας είναι μικρομεσαίες. Θα λειτουργήσει σε εθνική νομοθεσία που μπορεί να είναι πιο αυστηρή από την νομοθεσία που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. δεύτερη μου ερώτηση είναι ότι δεν υπάρχει ρήτρα που να διευκρινίζει ότι η εθνική νομοθεσία είναι καλύτερη για την μικρομεσαία ο προαιρετικός, η προαιρετική συμβατική νομοθεσία 88 ε, δεν θα ισχύει εφόσον τα δύο συμβαλόμενα μέρη έχουν ε, συμφωνήσει για να συνάψουν ευρωπαϊκό, ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Αυτά είναι σημαντικά θέματα και είμαστε διαθέσιμοι να συμμετέχουμε στα εργαστήρια που θα γίνουν από την, θα διοργανωθούν από την Επιτροπή Γιούρι. Αλλά αν σήμερα μπορούσατε κάπως να με ενημερώσετε για το πώς προτίθεστε να προετοιμάσετε αυτή την νομοθεσία και πώς θα εφαρμοστεί αυτή θα με βοηθούσε πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Όλσον. Εκπαιδευτική Ένωση ε, Κινήματος Ενυφαλιότητας. Εδώ βρίσκομαι για να με δείτε. Εγώ θέλω να ξέρω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Γίνεται πολλής λόγος για αυτή την ατζέντα που θα πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά και το σε βάλω τους ανθρώπους. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το αλκοόλ και για το κατά πόσο υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης για τα προϊόντα αυτά που ε, θα στο, σκέψετε το, τα εινοπνευματόδη και αν όχι γιατί όχι. Και τώρα ο κύριος Δελαλέ Τεστασά. Εγώ έχω μια ερώτηση που σχετίζεται με τα σημεία που υπάρχουν που αναφέρονται μέσα στο πρόγραμμα εργασίας 2012 της Κομισιόν που προβλέπει ένα μέσο για να αντιμετωπίσει το θέμα ε, των ε, δικαιωμάτων ασφάλισης. Ε, εκεί φαίνεται η Κομισιόν να προσανατολίζει ένα προαιρετικό μέσο. Εγώ σας έστειλα εδώ το Legislation and Welfare, μια, ένα, κατά τη γνώμη μας οι νομοθεσίες δεν έχουν στόχο μόνο την εναρμόνιση της εσωτερική αγοράς, αλλά και άλλες ε, ε, ανάγκες. Ο τομέα των ασφαλίσεων είναι πολύ ιδιαίτερος. Όπως γνωρίζετε, μέσω των ασφαλίσεων διοργανώνεται η ανάληψη των κινδύνων που σχετίζονται ε, με τη ζωή στην κοινωνία. Αυτή η δυνατότητα έχει εφαρμοστεί από πολλά κρατημένα. Για παράδειγμα, λαμβάνει κανείς, αναλαμβάνει μάλλον τις κινδύνους πλημμύρας σε ζώνες που μπορεί να πάσχουν από αυτό ή συλλειτουργεί ως μέσο κοινωνικής ασφάλισης επίσης και δεν θα πρέπει μια τέτοια νομοθεσία να σαρώσει όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες. Δεν υπάρχει χώρος, θα έλεγα, για προϊόντα τα οποία αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές λογικές, δηλαδή προϊόντα τα οποία θα είναι πολύ βαριά πλαισιωμένα, δηλαδή προϊόντα που αντιστοιχούν σε εθνική νομοθεσία ε, και πιο αμβλημένα στοιχεία ε, προϊόντα τα οποία αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκή νομοθεσία που προσπαθεί να βρει ένα κοινό παρονομαστή ανάμεσα στις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες αλλά που κατά κάποιο τρόπο θα παρέκαμπτε τις εθνικές νομοθεσίες. Θέλω λοιπόν να γνωρίζω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει το τι θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο μέσο και έχει ήδη αποφασίσει για μια νομοθετική μέθοδο. Θα ήθελα επίσης να σας δώσω τη θέση τη Ένωση μα για αυτό, Ένωσής για αυτό το θέμα. Εμείς πιστεύουμε ότι μια μήνυμο ε, ε, εναρμόνιση θα ήταν πιο κατάλληλη, που θα συμπληρώνεται από μια προσέγγιση προαιρετική, όπου θα τίθεται σε εφαρμογή κάποιες κοινέ αρχές, στι στις οποίες μάλλον θα καλούμε τον ε, κλάδο να προσχωρήσει. Ευχαριστώ. Κρίση Τζοβάνι από το Altro Consumo. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι εγγεγραμμένη για το, την τέταρτη συνεδρία για την επιβολή. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που να θέλουν να πάρουν το λόγο για... Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Όχι. Πολύ ωραία. Let uh, um, Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που Και η Πάολα Τεστόρη θα παρέμβει για ερωτήσεις που αφορούν το δικό της ε, τομέα. Για την ψηφιακή πτυχή της ε, ατζέντα του καταναλωτή. και λαμβάνοντα υπόψη την ψηφιακή πτυχή των πραγμάτων όταν νομοθετούμε. Αναφερθήκατε στην προστασία των δεδομένων. Και νομίζω πω όντω είναι πολύ κέρια αυτή η παρατήρηση, γιατί η Κομισιόν καταρχήν θέλει να φτιάξει ε, να στηρίξει μάλλον το οικονομικό ζήτημα της οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην ψηφιακή αγορά ε, ενισχύοντας ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών και αυτό το κάναμε ενισχύοντας το δικαίωμα να ξεχαστεί κανείς ενισχύοντας την κοινοποίηση δηλαδή περί των στοιχείων, ενισχύοντας επίση τη διαφάνεια για την πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τον καθένα. Έχουμε κάνει τεράστιε προσπάθειες για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και αυτό ισχύει ε, και για το να κάνουμε μια σύνδεση, γιατί έτσι οικοδομώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά ή στην τεχνολογία, ε, θα στηρίξουμε την ανάπτυξη. Αναφέρατε επίσης ότι Αναφέρεται βέβαια το γεγονός ότι όταν έχουμε πρόβλημα στην προστασία των ε, δεδομένων, τι θα κάνουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε. Εδώ θα ήθελα να τονίσω πως υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο στην προβλεπόμενη νομοθεσία που θεσπίζουμε αυτό που, λέμε, που ονομάζουμε αντιπροσωπευτική δράση. Γιατί λέμε συγκεκριμένα στην νομοθεσία ότι ο καταναλωτής το υποκείμενο των στοιχείων, όπως τον αποκαλούμε, μπορεί να στραφεί σε κάποια ένωση που ειδικεύεται στην προστασία των δεδομένων και αυτή η ένωση μπορεί να υπερασπιστεί την υπόθεση του εν λόγω καταναλωτή. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει στην θέσπιση αυτών των ε, προσωπικών δράσεων διότι διαπιστώνουμε πως όταν είσαι κανείς ε, ένα άτομο θα πρέπει να μπορεί ας πούμε να αγωνιστεί κατά της Google για παράδειγμα οπότε δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνος του το έχουμε λοιπόν αυτό σχεδιάσει συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές για την συντονισμένη προσέγγιση, το name and shame, που είναι ένα θέμα ε, το οποίο ε, έθεσε ο κύριος Τζούλ για το αν μπορούμε να διευκολύνουμε τα πράγματα για τους κατανοητές και να τους βοηθήσουμε στο να εντοπίσουν τις παγίδες, τις δυσκολίες που μπορεί κανείς να συναντήσει αντί να χρειαστεί να πάνε στο, στα δικαστήρια. Εδώ θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Πάολα γιατί αυτή είναι η δράση της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ για να βοηθηθούν οι καταναλωτές και να μπορούν να δείξουν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό στον τομέα των ε, χρηματοπιστωτικό. Είναι ένας ε, τομέας που εσείς αναφέρετε, αλλά ίσως εσύ Πάολα να μπορούσες εδώ να πεις δύο λόγια παραπάνω. Ευχαριστώ. Όπως είπα και νωρίτερα, στη ΣΑΝΚΟ συνεργαζόμαστε με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών αλλά και με τις οργανώσεις καταναλωτών που βοηθούν τους καταναλωτές και σε εθνικό επίπεδο και χρηματοδοτούμε τα δίκτυα αυτά του ECC και στο νέο πρόγραμμα, όπως είπα, αυξάνουμε μάλιστα την ε, χρηματοδότησή μας το 70% γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι σε όλες τις χώρες μέλη υπάρχει ένα μέρος όπου οι καταναλωτές και οι οργανώσεις καταναλωτών μπορούν να πάνε για να ζητήσουν συμβουλές. Τώρα για τον Οικονομικό Σύμβουλο, που είναι ένα σημαντικό θέμα και εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ξέρουμε ότι ζητήσατε ένα εκατομμύριο για να χρηματοδοτηθεί αυτή η Οικονομική Συμβουλή. Τι σημαίνει, σημαίνει ανεξάρτητη βέβαια συμβουλή, έτσι, δηλαδή τράπεζες ή τα δημοσιονομικά όργανα Μπορούν να είναι ένας ανεξάρτητος σύμβουλος. Κατά πάσα πιθανότητα η απάντηση είναι όχι. Οπότε εμεί θέλουμε να ενισχύσουμε μονάδες σε εθνικό επίπεδο που να μπορούν να συμβουλέψουν οικονομικά τον καταναλώτη. Αλλά για να γίνει αυτό οργανώνουμε και μια κατάρτιση. Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα. Κάτι άλλο που είπατε είχε να κάνει με την άλκο. Συγγνώμη, έχει να κάνει με τα ενοπνευματόδη. Προκειμένου ε, πώς θα μειωθεί η κατανάλωση νοπνεύματος από τους νέους. Εμείς στα κράτη-μέλη, εκεί που εμείς συντονίζουμε την δράση των χωρών μελών, για την πώληση, για παράδειγμα, υπάρχει περιορισμός ε, όσον αφορά τις αρμοδιότητές μας. Πιέζουμε όμως και συντονίζουμε τη δράση των χωρών μελών. Και δεύτερον, έχουμε και μία πλατφόρμα όπου συνεργαζόμαστε με τη βιομηχανία και πιέζουμε τη βιομηχανία να υιοθετήσει ένα κώδικα δεντολογίας και έναν ε, περιορισμό διάθεσης στην αγορά. Γιατί βλέπετε το πρόβλημα της κατανάλωσης ε, αλκοόλ ε, με τους νέους περνάει και από εκεί. Γι' αυτό και θέλουμε προαιρετικά την συνεργασία της βιομηχανίας. Δουλεύουμε λοιπόν και πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Πάολα. Τέλος, για το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων, που ρωτήσατε, έτσι δεν είναι. Ή... Α, και μετά θα σας δώσω το λόγο, θα σας δώσω το λόγο μετά. Έλεγα λοιπόν και το ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εδώ να υπογραμμίσουμε ότι σχεδιάζοντας ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων, όπως κάναμε και με την προστασία δεδομένων, προσέξαμε όλος ιδιαιτέρως το 99,9% των επιχειρήσεων που είναι τελικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το κοινό δίκαιο πολίσεων είναι κάτι από το οποίο έχουν να επωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα υπάρξει μεγάλη απλοποίηση ώστε να έχουμε το ίδιο σύστημα εφόσον υιοθετηθεί σε όλες τις χώρες μέλη. Αναφερθήκατε στην περίπτωση της σχέσης μιας μεγάλης επιχείρησης με τις μικρομεσαίες. Υποθέτω ότι θέλετε να πείτε πως αυτό το δεύτερο καθεστώς μπορεί να επιβληθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, είναι μια γενική προβληματική που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγώ ασχολούμαι τα τελευταία πέντε χρόνια με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ξέρω ότι μερικές φορές βρίσκονται σε δύσκολη θέση. όταν βρίσκονται αντιμέτωπε με μια μεγάλη επιχείρηση. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και είμαστε έτοιμοι να δούμε υπό το πνεύμα του στόχου μας που είναι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κάτι που και πρόσφατα έχει επιβεβαιώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν παρετέρω στα πλαίσια των συζητήσεων αυτών που θα λάβουν χώρα στη συνέχεια. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε με το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων, όπω και με οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία, είναι να εποφελούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Τέλο για την, ε, τις ασφάλειες. Για τι ασφάλειε, είμαστε σε μια κατάσταση όπου προβληματιζόμαστε. Θα έχουμε διαβούλευση με τον κλάδο, θα μελετήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε πριν να καταλήξουμε σε κάποια κατεύθυνση, πόσο μάλλον σε συμπεράσματα. Έχουμε επαφές με τον κλάδο και θα συνεχιστούν. τα τη διάρκεια του 2012 θα συνεχιστούν αυτές οι επαφές για να καταλήξουμε στο τι τελικά χρειάζεται στον τομέα αυτό της οικονομίας. Άρα προς το παρόν δεν υπάρχει κατεύθυνση. Η κυρία Ριγόνια, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα έχω να κάνω και εγώ κάποια σχόλια με τα από όσα άκουσα. Φυσικά και θέλω να επιθυμίσω, γιατί το ξεχνάμε συχνά, ότι όλοι είμαστε καταναλωτές, πολίτες. Άρα έχουμε κάποια δικαιώματα, έτσι κι αλλιώς. Τι θέλει ο καταναλωτής και οργανώσεις καταναλωτών από τον ε, νομοθέτη, προστασία και πρόληψη. Γιατί για να είμαστε μοιημένοι και ενημερωμένοι καταναλωτές, αυτό χρειάζεται. Κάποιος μίλησε για ευφυείς μάλιστα καταναλωτές. Ε, μακάρι κάποια στιγμή να είμαστε όλοι ευφυείς καταναλωτές. Οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν ή να μην ζητήσουν αποζημίωση. Πρέπει όμως να έχουν το δικαίωμα, γιατί αν θέλουν να ζητήσουν την αποζημίωση, ακόμα και αν είναι για 10 ευρώ, πρέπει να έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Έπειτα η κρίση δεν μειώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αντίθετα τα ενισχύει. Ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση των ευάλωτων καταναλωτών που δεν πρόκειται μόνο για την ενημέρωση, πρόκειται για πολύ περισσότερα πράγματα και αυτό πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Ριγόγεν. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ. Μήπω έχουν επιπλέον σχόλια. I've got one comment in relation to... Uh, ναι, εγώ έχω ένα σχόλιο όσον αφορά την προστασία των ε, δεδομένων και την σχέση μεταξύ προστασία δεδομένων και προστασία καταναλωτή. Υπάρχουν δύο πτυχέ. Η μία είναι εκεί όπου οι καταναλωτέ ε, δίνουν ε, με τη θέλησή του τα δικά του προσωπικά στοιχεία ε, εδώ ε, πρόκειται για ένα πράγμα το οποίο έχει οικονομική αξία. Τα αγαθά έχουν οικονομική, τα στοιχεία έχουν οικονομική αξία. Ο καταναλωτή όμω δεν το καταλαβαίνει πάντοτε αυτό. Άρα ο καταναλωτή θα έπρεπε να μπορεί να πουλήσει τα προσωπικά του δεδομένα. Να αποζημιώνεται με κάποιο τρόπο. Να έχει κάποιο όφελος όταν δίνει τα στοιχεία του οι καταναλωτέ, όταν, παίρνουν, όταν τα στοιχεία του τους ε, τα δίνουν ε, σιωπηρά ή ε, κρυφά χάνουν ε, κάποιο δικαίωμα σε αποζημίωση. Μια από τι δυσκολίε λοιπόν που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με συνεργασία με άλλε αρχέ επιβολή εντό και εκτό τη ε, Ένωση σχετίζονται με του κανόνε προστασία δεδομένων που υπάρχουν για καλού λόγου, αλλά το αρνητικό είναι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να έχουμε βάση δεδομένων για τι καταγγελίε των καταναλωτών και άρα και πλήρη εικόνα για το τι ακριβώ συμβαίνει εντό και εκτό Ένωση. Για τι αγγλόφωνε χώρε είναι ιδιαίτερα προβληματικό, ακόμα και αν η ίδια επιχείρηση που λειτουργεί ας πούμε στο ΕΠΑ, λειτουργεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο και θέλουμε να έχουμε πλήρη εικόνα, αλλά είναι πολύ δύσκολο λόγω των διαφορών που υπάρχουν στην προστασία των δεδομένων ε, να μοιραστούμε τα στοιχεία με τους Αμερικανούς συναδέλφους. Γι' αυτό νομίζω πρέπει αυτό το θέμα να διεξεταστεί περαιτέρω. Σας ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνέδρους για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, συμβολές τους. Σας ευχαριστώ όλους. thank Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που συντονίσατε αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης και τώρα θα περάσουμε στη τρίτη συνεδρία. Κάπως έχουμε μείνει πίσω. Ε, ζητώ συγγνώμη που σας πιέζω κάπως τους ομιλητές, αλλά ελπίζω πως θα έχουμε και χρόνο για συζήτηση. Εδώ έχουμε πολλούς ομιλητές ε, και πάλι από το ακροτήριο. Αν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις ε, στον τομέα της ενημέρωσης και της παιδείας, θα δώσω το λόγο ήδη στον συντονιστή, στον David. So I'm very pleased um, to welcome um, uh, someone who I can say is a long-standing friend. Να καλωσορίσω έναν παλιό φίλο της, Επιτρο... της Επιτροπής μας, um, και ε, που έχει συνεισφέρει στην εργασία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και τον καλωσορίζω πρώτη φορά στην, υπό τη νέα του ιδιότητα, που, καθώς εργάζεται για το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως επικεφαλής της μονάδας για τις επιστήμες, τι τις επιστημονικές συμβουλές για την πολιτική. Δίνει πολλά σημαντικά στοιχεία που εμείς χρησιμοποιούμε, ιδιαίτερα το πίνακα επιδόσεων των καταναλωτών και το πίνακα επιδόσεων της αγοράς που μας βοηθούν να καταλάβουμε τη λειτουργία των αγορών. Και νομίζω πως η παρουσίαση του κυρίου Φρήμαν, με την οποία συμφωνώ απόλυτα, υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο το πώς λειτουργούν οι αγορές για να μπορέσουμε να προστατέψουμε. Το, αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε και με τον κύριο Αλμούνια. Αυτά λοιπόν. Μια γενική είπα, λοιπόν εισήγηση από μένα ως πρόεδρο και να δώσω το λόγο στον David Μέρ που θα είναι και ο συντονιστής της επόμενης συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ Μάλκομ, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Για όσους δεν γνωρίζετε το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, να πω ότι είμαστε το η Εσωτερική Επιστημονική Υπηρεσία της Επιτροπής. Θέλουμε να, έργο μας είναι να προσφέρουμε επιστημονική σύμβουλη επιστημονικέ συμβουλέ και να βοηθήσουμε την Κομισιόν να προωθήσει τις, και να σχηματίσει τι πολιτικέ τη. Τα τελευταία 13 χρόνια εργαζόμουν για την πολιτική του καταναλωτή στην, Επιτροπή, στην ε, διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και εξακολουθώ να ενδιαφέρομαι για αυτά τα θέματα, ακόμα και αν τώρα εργάζομαι σε διαφορετικό τμήμα της Επιτροπής, γιατί η ενημέρωση και η παιδεία είναι τόσο σημαντικές. Φυσικά και είναι σημαντικές για την ευημερία των καταναλωτών, για να μπορούν να προβαίνουν σε ε, ε, σωστές επιλογές, πράγμα το οποίο είναι θεμελιώδες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία. Πολύ καλή δουλειά έκαναν όσοι κέρδισαν το Nobel Prize για την οικονομία πέρυσι, όπου ανακάλυψαν το παράδοξο του διαμαντιού, όπως αποκλήθηκε. Δηλαδή ότι στις αγορές όπου τα αρχικά κόστη είναι πολύ ψηλά, που σημαίνει δηλαδή ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν εύκολα να υπολογίσουν την τιμή και αν είναι ψηλή ή χαμηλή. Σε αυτές τις αγορές, ακόμα και αν υπάρχουν πολλοί φορείς και φαίνεται να είναι πολύ αντιγωνιστικοί, αυτές οι αγορές αρχίζουν και συμπεριφέρονται ως μονοπόλια. Αν λοιπόν οι καταναλωτέ δεν μπορούν ενημερωμένα να προβούν σε επιλογέ για το ποια είναι καλύτερα, τα καλύτερα προϊόντα και η καλύτερη σχέση ε, με την τιμή και ποια είναι η καλύτερη εταιρεία με την οποία μπορούν να συνεργαστούν, τότε οι αγορέ αυτέ αρχίζουν να μοιάζουν με μονοπωλιακέ αγορές. Φαίνεται να έχουν παίκτε πολλού, να συμμετέχουν πολλοί παίκτε, αλλά επειδή είναι τόσο δύσκολο να βρει κανεί το καλύτερο προϊόν, φαίνεται να μην είναι σωστέ και ανταγωνιστικές. Η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει ο καταναλωτή αυτή τη στιγμή δεν είναι στατική. Είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση και μεταβαλλόμενη. Υπάρχει υπερβαλλικός φόρτος προσφοράς, ο αριθμός των προϊόντων που είναι υποπόληση, η εξάπλωση των σημάτων, ο πολλαπλασιασμός των λογοτύπων και ούτω καθεξής. Αυτό που βλέπουμε μέσω των ε, επιστημών συμπεριφοράς είναι ότι όλα τα άτομα και οι καταναλωτές έχουν συγκεκριμένους γνωστικούς περιορισμούς όσον αφορά την κατανόηση και την επιλογή. Και αυτό είναι κάτι που συστηματικά ισχύει για... και το αναγνωρίζουν όλοι όσοι εργάζονται στους εκπαιδευτικούς τομείς. Επίσης αυτό που βλέπουμε είναι πως στους δυναμικούς τομείς οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν αυτούς τους ε, γνωστικούς περιορισμούς και οι διαφημίσεις γίνονται όλο ένα και πιο προηγμένες και προσαρμόζονται στους γνωστικούς περιορισμούς των καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά όμως είδαμε τελευταία μέσω της ανάπτυξης του Ιντερνετ μια ε, τεράστια αύξηση σε, των νέων ενδιάμεσων που διευκολύνουν τους καταναλωτές να προβούν στις σωστές επιλογές και κατά τη γνώμη μου αυτό προσφέρει τεράστιες ελπίδες ώστε να μπορέσουν οι καταναλωτές να βρουν το δρόμο τους μέσω των δύσκολων και περίπλοκων επιλογών που αντιμετωπίζουν όλο ένα και περισσότερο. Να μπορούν δηλαδή να προβαίνουν στις επιλογές που χρειάζεται για τον εαυτό τους αλλά και για να μπορεί η αγορά να λειτουργεί σωστά και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Έχουμε τρεις πολύ καλούς ομιλητές σήμερα το πρωί για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Πρώτα έχουμε τον Λούι Γκρέχ που εκτό που είναι αντιπρόεδρο τη επιτροπή ε, ΙΜΚΟ ήταν και εισηγητή τη πολύ σημαντική έκθεση για την ενιαία αγορά και του πολίτε. Και νομίζω ότι είναι ο άνθρωπο που καταρχήν ε, έφτασε στην φανταστική ιδέα για το ποια είναι τα 20 πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτε στην ευρωπαϊκή αγορά. Και αυτό απογειώθηκε ω ιδέα και έχει μετατραπεί σε πολύ σημαντική βάση. Έπειτα έχουμε τη Μονίκο Γιένς, που είναι γενικός, γενική διευθύντρια τη ΜΠΕΟΚ, και τέλος ο συνάδελφος Τζεραρ Ντεγκράφ, που είναι διευθυντής στην ε, Γενική Διεύθυνση ΙΜΣΟ για τα οπτικοακουστικά μέσα και την πολιτική ενημέρωση, αλλά και για τις ηλεκτρονικέ επικοινωνίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Λουι Γκρέγνα που θα μας πει δύο λόγια για την έκθεση που συνέταξε για την νέα αγορά και τους πολίτες. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα κάπως σύντομα να επικεντρωθώ στο τι τελικά ε, προσφέρουμε με την εσωτερική αγορά προς τους πολίτες μας, τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πριν από μισό χρόνο είχα πει ότι χρειαζόμασταν ε, μια συνολική σφαιρική στρατηγική η οποία να επικεντρώνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της αγοράς. Όπως αναγνωρίζω και στην έκθεσή μου, η ενεργός συμμετοχή των καταναλωτών στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί ο κάθε καταναλωτής βλέπει διαφορετικά, ας που δεν ασχολείται και πολύ με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Έπειτα, η αντίληψη των καταναλωτών για την εσωτερική αγορά δεν έχει βελτιωθεί και πολύ τα τελευταία χρόνια. Για τους καταναλωτές λοιπόν η ενημέρωση αποτελεί μέρος διαπαιδαγώγησης. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια στρατηγική για την ενημέρωση ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη σωστή ενημέρωση και να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν εν γνώση του τι κάνουν. Επιμένω λοιπόν και ζητάω μία χάρτα δικαιωμάτων των πολιτών που θα υπογρομίζει και τις υποχρεώσεις των πολιτών στην ενία αγορά με έναν εύκολα κατανοητό τρόπο. Πρόεδρε, η Επιτροπή ΙΜΚΟ συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αυτή. Φυσικά δεν μπορούμε εδώ πέρα να καλύψουμε όλες τις πτυχές του έργου της ΣΥΜΚΟ. Παρόλο έχουμε προτείνει διάφορα μέτρα νομοθετικά και μη για την πολιτική υπέρ των ε, πολιτών. Για παράδειγμα την ε, ε, πράξη για την ενιαία αγορά, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την μελέτη για το 2020. Επιπλέον, η Επιτροπή και ιδιαίτερα η Επίτροπη Δαλή και Ρέντινγκ ανταποκρίνονται και επικεντρώνονται στις ανησυχίες των πολιτών προτείνοντας την ε, αναθεώρηση ε, και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, οδηγίες και κυρίως το θέμα των εναλλακτικών ε, επιλύσεων διαφοράς. Όλα αυτά φάνηκαν και στην μελέτη για το 2020. Πρώτα απ' όλα φαίνεται από εκεί η απογοήτευση των πολιτών απέναντι στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν και ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει καλές λύσεις για τα 20 προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Επιπλέον, λαμβάνοντα υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν εντοπίσει τι ελλείψει και τι αδυναμίε τη αγορά και έχουν εγκρίνει κάποια αναγκαία νομοθετικά μέτρα, τώρα πρέπει να περάσουμε στο πιο σημαντικό στάδιο και αυτό είναι ενιαία αγορά που οι διατάξεις της να εφαρμόζονται και να γίνονται αποδεκτές από όλες τις χώρες μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτό το τρίτο στάδιο πανεκκίνησης της εσωτερικής αγοράς. Φυσικά θέλουμε και μια αναθεώρηση στα μέσα του δρόμου για να δούμε ο χάρτης αυτός πορείας έχει πετύχει τους στόχους του. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στην ΕΜΚΟ και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές μια τέτοια αξιολόγηση εφόσον την έχει. Τέλος, η εσωτερική αγορά είναι 20 ετών μπορεί να αποτελέσει καταλητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας, προστατεύοντας συγχρόνως τον καταναλωτή. Η κρίση είναι σοβαρή. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Παραμένουν σημαντικές προκλήσεις μπροστά μας. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι κάτι που μπορεί να πάει πίσω και είναι ευθύνη των χωρών μελών να νιώσουν ότι ανήκουν σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι δικιά τους να την ιδιοποιηθούν και έτσι να προχωρήσουν στην στήριξη της εσωτερικής αγοράς. Αν δεν δώσουμε αποτελέσματα στους πολίτες, οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εγκαταλείψουν την όλη διαδικασία, η οποία θα πάει προς τα πίσω αντί να πηγαίνει μπροστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε γρήγορα. Μονίκο Εν, επόμενο μιλείτε, για να μας πείτε τη δυνατότητα δημιουργίας ε, δυναμικού και τη ρόλου του ε, συνηγόρου του καταναλωτή. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω κάποια γενικά πράγματα καταρχήν, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι εμεί από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την ανακοίνωση που έκανε η Κομισιόν για την προετοιμασία μια ατζέντα για τον καταναλωτή, παρόλο που δεν ξέρουμε ακόμα το περιεχόμενο τη, που θα ήταν το πιο σημαντικό για μα. Πιστεύουμε επίση ότι δίνεται ένα πολύ έντονο μήνυμα προ του καταναλωτέ τη Ευρώπη ότι θα είναι στο επίκεντρο τη ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το, οι απαντήσει στο feedback που έχουμε από τα μέλη μα είναι ότι η ενιαία αγορά είναι πολύ μερικό επίτευγμα η πράξη για την νέα αγορά αντιμετώπισε κάποια από τα θέματα, αλλά εξακολουθούν από σκοπιά καταναλωτή να υπάρχουν πολλά κενά. Επίσης ε, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι για την ευμάρεια του καταναλωτή χρειάζεται πολύ περισσότερο από ότι μόνο ε, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η ευημερία του εξαρτάται και από άλλους παράγοντες θα έχουμε ένα έγγραφο πρόσεγό και θα το δώσουμε στα θεσμικά τη ημέρα και σε μερικέ εβδομάδε πιο ευρέω. Όπω ο Επίτροπο Δαλή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση. Δεν είναι πρώτο δηλαδή, το θέμα, δηλαδή μόνο για τα δικαιώματα των καναλωτών περιορισμένα, είναι το θέμα τη απελευθέρωση των ε, ε, αγορών ενέργεια, αποτελεσματική χρήση τη ε, ενέργεια, μεταφορέ κλπ ότι έχουν ε, για την προετοιμασία της ακρόασης αυτής και ακούγοντας τα πρώτα που ελέγξαν, ε, είχα πραγματικά πολλές ανησυχίες αρχικά. Είχα την εντύπωση ότι πρόκειται για ε, τίτλους ε, κλασικούς προστασίας του κατανοητή Δηλαδή ασφάλεια, πληροφόρηση, ενημέρωση κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει όμως μια νέα προσέγγιση. Και φάνηκε αυτό και από τη συζήτηση. Με καθυστέρηση, καθυσ σύχασαν δηλαδή αυτά που είπε ο Επίτροπος Νταλή που είπε ότι και εκείνο ε, έχει κάπως συγχυστεί γιατί δεν καταλαβαίνει πολύ καλά τη σχέση μεταξύ της ε, στρατηγικής για τον καταναλωτή και της, ε, και της πρόθεσης του καταναλωτή. Και μετά ανησύχησε γιατί είπε ο ο κύριος Νταλή ότι το πρόγραμμα για τον καταναλωτή θα είναι η οικονομική ε, ερμηνεία, αν θέλετε, της ε, ατζέντα για τον καταναλωτή. Αλλά αυτό με ενίσχυσε πάρα πολύ γιατί ε, έχουμε την σάκο εδώ, άρα δεν έχουμε μόνο σφαιρική προσέγγιση, έχουμε και κάτι παραπάνω. Ακούσαμε διάφορα όσον αφορά για την αρμοδιότητε που πρέπει να δοθούν στην ε, καταναλωτή. και έχω εμπιστοσύνη ότι ο Επίτροπος Δαλή και οι υπηρεσίε του ξέρουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ φιλόδοξη προσέγγιση είδα σε πολλούς τομείς ότι αυτό σημαίνει απλώς να του ρίχνουν κάποιες πληροφορίες του καταναλωτή χωρίς ε, να ξέρει τι να τις κάνει. Και η ευθύνη μετά μεταβιβάζεται στον καταναλωτή αν δεν πάρει σωστές αποφάσεις. Το είπε και ο κύριος Φρήμαν. Θα πρέπει να έχουν τα μέσα οι καταναλωτές για να κάνουν τις σωστέ επιλογές. Ο Ντέιβιτ είπε ότι το διαδίκτυο έχει ένα τεράστιο δομικό να δώσει ε, δικαιώματα στου κατανοητέ για τι επιλογέ που μπορούν να κάνουν. Από την άλλη μεριά όμως ενέχεται και πάρα πολλού κινδύνους που δεν υπήρχαν στο παρελθόν γιατί δεν υπάρχει επικύρωση των ε, πληροφοριών όπω α πούμε αυτό το σκάνδαλο για του συμβούλου για το TRIP και μετά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και πολλέ αντιφατικέ πληροφορίε. Και είδαμε τελικά ότι οι καταναλωτέ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τι αντιφατικέ ε, πληροφορίε και αυτό δεν ισχύει μόνο στην βιομηχανία αλλά και στι δημόσιε αρχέ. Ε, δείτε, α πούμε, όσον αφορά αυτά τα. αυτό το πρόβλημα με τα εμφυτεύματα ε, μαστών που η Ισπανική κυβέρνηση είπε στους καταναλώτες ότι δεν πειράζει να τα κρατήσουν, η Γαλλική είπε πρέπει οπωσδήποτε να τα βγάλουν. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να ενημερώνεται και να εκπροσωπείται σωστά ο καταναλωτής. Και αυτό πήρα, ένα λεπτό από τον, από τον συνάδελφο εδώ. Συμφωνεί. Καλή συνεργασία αυτή για να μπορεί ε, να είναι κανένας αξιόπιστη οργάνωση των καταναλωτών σημαίνει ότι πρέπει να έχει επίτρεση στους νομοθέτες, να έχει συνεργασία της με την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια συνεχόμενη πρόκληση και πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να το κάνουμε. Αυτό είναι μια πρόκληση για όλες τις οργανώσεις των καταναλωτών στην Ευρώπη και έχει δραματική θετική εικόνα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όπου η πολιτική για τους κατανοητές βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα και δεν υπάρχει αυτή η παράδοση, η οργανώση των καταναλωτών να είναι αξιόπιστη ε, εταίρη των κυβερνήσεων. Αναγνωρίσαμε τις ε, δυσκολίες, χρηματοδοτήθηκαν οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους καταναλωτές και τους έδωσαν πολλές δυνατότητες. Είναι νομίζω κρίσιμο να συνεχίσουμε χιστεί η ίδια κατεύθυνση και ε, με σίγουρο θα να κοινωθεί κάτι τέτοιο, αλλά παρακαλώ η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα να έχουν επίδραση στα κράτη-μέλη, στι κυβερνήσει του εκείνοι να αρχίσουν να ακούνε τι οργανώσει των καταναλωτών. Ακόμη και στι χώρε που δεν υπάρχει παράδοση για κάτι τέτοιο. Monique, uh... Ε, Ευχαριστώ πολύ, Μονίκ. Τζεραντ, ευκαιρίε και κίνδυνοι ενδεχομένω τη ε, ψηφιακή κοινωνία. Δύο λεπτά έχω στη διάθεσή μου, οπότε θα μιλήσω όσο πιο γρήγορα μπορώ και θα περιοριστώ στα σχολιά μου βέβαια. Δεν θα κάνω καμία εισαγωγή. Πρώτα απ' όλα, ο ανταγωνισμό είναι πάρα πολύ καλό για του καταναλωτέ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ιδιαίτερα στι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε έχουμε απόδειξη γι' αυτό. Έχουν μειωθεί οι τιμέ, έχει αυξηθεί η επιλογή. Πολύ καλά όλα αυτά. Οι αγορέ δεν είναι τέλειε. Το έχουμε δει αυτό και στι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε. Το ξέρουμε με το roaming, για παράδειγμα, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν ε, καλό που έχει μειωθεί κατά 70% από το 2007 η τιμή και θα υπάρξουν και άλλες παρατέρω Πολύ καλό αυτό. Είναι ένα επίτευγμα. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι η εσωτερική αγορά στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ο κύριος Γκρέκ το είπε στο δικό μας τον τομέα είναι αλήθεια αυτό. Ακόμα έχουμε πολλά να κάνουμε, να εξακολουθήσουμε να μελετάμε και θα το κάνουμε στα τελευταία του μήνα ε, τις τιμές των ε, μη ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών ε, επικοινωνιών. Για την ενημέρωση τώρα και τη διαπαιδαγώγηση του κοινού. Πρώτα απ' όλα, αν οι καταναλωτέ δεν γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα για τα δικαιώματά του Και ένα από τα πράγματα που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να δημοσιεύσει έναν κώδικα για τα δικαιώματα online. Πολύ καλό αυτό για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι δικαιώματα έχουν και πώ είναι προστατευμένοι. Καλύτερη ενημέρωση λοιπόν, όχι περισσότερη, καλύτερη. Γιατί έτσι αυξάνει και η εμπιστοσύνη. όπω όμω είπε και David, είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία και των αγορών η ενημέρωση. Ένας τώρα από τους τομείς που εξετάζουμε εμείς στενά είναι πώς γνωρίζουν οι καταναλωτές μας τι παίρνουν ε, στο διαδίκτυο σταχύτητα. Πολλές φορές ε, γράφεσαι για 30 MB και παίρνεις 10. Η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές δεν ξέρουν πάντα αν παίρνουν αυτό για το οποίο πληρώνουν και αν δεν το παίρνουν να μπορούν να αλλάξουν. Αυτό πρέπει να υπάρχει. Είναι μια διαφάνεια και αυτή που πρέπει να έχουν οι καταναλωτές και το δικαίωμα να μπορούν να αλλάζουν. 26 δευτερόλεπτα κέρδισα από το χρόνο μου, οπότε σταματάω εδώ, λέει ο κύριος Ντεχράφ. Ευχαριστούμε πολύ, Γκέραρτ. Τέσσερις έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν θα προφέρω καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πρώτα έχω την κυρία Ροτσίτσκα, από την οργάνωση Πολωνών Καταναλωτών είναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Θα ξεκινήσω με κάτι θετικό. Η ιδέα του να έχουμε έναν ισχυρό καταναλωτή στο κέντρο της εσωτερικής αγοράς είναι πολύ θετικό. Επίσης, είναι θετικά και τα επιτεύγματα που έχουμε μέχρι τώρα στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών. Όμως, ο στόχος μας που είναι να είναι ο καταναλωτής στο κέντρο της εσωτερικής αγοράς είναι κάτι που πρέπει να φροντίζουν οι οργανώσεις καταναλωτών. Βλέπετε η πραγματικότητα είναι τέτοια που πολλές οργανώσεις καταναλωτών περιορίζουν τις δυνατότητες δράσης και λειτουργίες τους. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με την οικονομική κρίση σε έναν βαθμό, αλλά επίσης επειδή πολλές τέτοιες οργανώσεις λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες στις χώρες τους, οπότε δεν έχουν πολλές δυνατότητες να επηρεάζουν την πολιτική και έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες να προωθήσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών με εργασίες ε, και ε, πρόθεση ιδεών στα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι ιδιαίτερα προβληματική. Όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε τις οργανώσεις των καταναλωτών, όμως πρέπει να αντιληφθούμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσουν. Περιμένουμε από αυτούς να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις και να φροντίσουν να είναι ανεπίτροπτη αυτή η απαγόρευση των οργανώσεων των καταναλωτών. Αλλιώς ποιος θα φροντίσει για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ευχαριστούμε. κούτιν τώρα, Σλοβενία, από την Σλοβενική Οργάνωση Καταναλωτών. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα συνεχίσω κι εγώ μιλώντας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εξακολουθούν να μας θεωρούν νέες χώρες μέλη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, οικονομικά μιλώντας και από πλευράς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Δυστυχώς ακούμε ότι πολλές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση του καταναλωτή είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Τα ακούσατε τι ισχύει σε πολλές χώρες αν λοιπόν θέλετε να ενισχύσετε τον καταναλωτή και να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη του στα καταναλωτικά προϊόντα, φυσικά και η ενημέρωση είναι πρωταρχικός παράγοντας σε μερικές ε, περιπτώσεις, λίγες, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα ε, μοιημένος να κάνει επιλογές μετά από συγκριτικές δοκιμές. Οι συγκριτικές δοκιμές ε, βελτιώνουν τη διαφάνεια, ευνοούν τις επιλογές του καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και εκείνη της ενημέρωσης κατά πόσο θα ήταν δυνατόν να στηρίξετε προγράμματα προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Δηλαδή να γίνονται μελέτες ώστε και να ενισχύεται ο καταναλωτής μέσω των οργανώσεών του ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε σε εθνικό επίπεδο συγκριτικές δοκιμές των προϊόντων. Ακούμε συχνά για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ναι, αλλά πώς θα το αποδείξουμε αυτό, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν λοιπόν θέλουμε διασυνοριακά οι καταναλωτές να αγοράζουν, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τέτοιες συγκριτικές δοκιμές στα προϊόντα. Αντινάσκομ από το φόκους των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ, εδώ είμαι. Ο Επίτροπος Νταλή ανέφερε νωρίτερα πόσο μεγάλη σημασία έχει το feedback, ε, τα σχόλια από τις οργανώσεις των καταναλωτών για να ξέρουν ε, τι πιστεύει ο καταναλωτής. Γι' αυτό και έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την κυρία Κογέννης για την ενεργειακή πολιτική. Για την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ που ε, συντονίζει κάπως ε, αυτό το input των καταναλωτών. Ρωτάω λοιπόν, μπορεί αυτό να επεκταθεί και σε άλλους τομείς πολιτικής. Τη Μονίκ θέλω να τη ρωτήσω το εξή. Είμαστε στα πέντε χρόνια του Φόρουμ των Καταναλωτών. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος διάλογος του φόρουμ αυτού με εθνικές οργανώσεις καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τέλος, στον κατάλογο μιλητών έχω την κυρία Σούλτου από το CCIR. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Unisol τον ονομάζομαι και εκπροσωπώ τους Ευρωπαίους ρυθμιστές ενέργειας και θέλω να έρθω σε αυτό που είπε και Χάιντι λιγάκι. Στον τομέα της ενέργειας πράγματι έχουμε ένα ετήσιο φόρουμ που ονομάζεται London Forum για τους καταναλωτές και ασχολείται με το θέμα ενέργειας και καταναλωτών. Εμείς προσωπούμε τους εθνικούς ρυθμιστές, το σώμα μας δηλαδή τους εκπροσωπεί και βλέπουμε τα δικαιώματά τους πώς αντιμετωπίζονται στο τρίτο πακέτο. Την τελευταία φορά που είχαμε δηλαδή νομοθεσία. Τώρα προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας την άποψη των καταναλωτών για το 2020. Δηλαδή η αγορά ενέργειας, η ευρωπαϊκή, τι πρέπει να δίνει στους καταναλωτές. Δεν προσπαθούμε εμεί δηλαδή να πούμε σε αυτού τι πρέπει να κάνουν, αλλά περιμένουμε να υπάρχει διάλογο με του καταναλωτέ μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμμετοχή όλων των διαφερομένων είναι κεντρική σημασία και μεγάλη βέβαια πρόκληση για μας είναι πώς θα ακούσουμε τη γνώμη του απλού πολίτη. Γι' αυτό και ρωτάω και τον κύριο Κρέκ να με συμβουλέψει. Πώς πιστεύει ότι μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορούμε να φτάσουμε στην εκλογική σας περιφέρεια για παράδειγμα, για να δούμε πώς βλέπουν οι καταναλωτές εκεί την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην τους βλέπουμε μόνο μία φορά το χρόνο στο φόρουμ του Λονδίνου και μόνο μία φορά το χρόνο να ακούμε από τις οργανώσεις καταναλωτών την άποψή του Ακούσαμε πολλές ερωτήσεις. Πρώτα η DG Sanko και μετά οι υπόλοιποι. Για να απαντήσω στη Μονίκη Κογκογιές. Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα για τον καταναλωτών καλύπτει ένα μέρος του προγράμματος για τους καταναλωτές της ατζέντα αυτής είναι όπως το είπα και πριν. Θέλουμε, ο Επίτροπος Ντάλι και Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ το λένε ότι η ατζέντα αυτή των καταναλωτών θέλουμε να καλύψει ολό, όλες τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές. Το θέμα είναι βέβαια οικονομική πόρη, έτσι και δεν ξέρω και αν ε, και οι άλλοι επίτροποι είναι τόσο πρόθυμοι όσο και εμείς να ξοδέψουν για τη στήριξη των καταναλωτών. Τώρα, δεύτερον, γιατί δεν κάνουμε περισσότερες δοκιμές προϊόντων στην αγορά. Κάνουμε μερικές. Το είπε αυτό και ο συνάδελφος από το POSAVE. Έχει να κάνει με την εποπτεία της αγοράς. Πάλι λέω ότι ο προπολογισμό είναι περιορισμένο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρηματοδοτούμε συντονισμένη δράση. Αλλά να πούμε ότι στην κάθε εθνική αγορά θα χρηματοδοτήσουμε τη δοκιμή προϊόντων, όχι, δεν είναι αυτό δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο. Πώ να έχουμε τη συμμετοχή του καταναλωτή στην εκπόνηση πολιτική. Όπως λέτε και εσείς στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και νομίζω ότι και πάλι Ακριβώς γι' αυτό είμαστε εδώ για να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Υπάρχουν και ένα βέβαια όσον αφορά τη διαβούλευση με ε, τους ενδιαφερόμενους. Αλλά το κανόνα του να θέλουμε αυτή την επαφή τον εφαρμόζουν και όλοι οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ Πάολο. Κύριος Γκρέκ ίσως για να απαντήσει για την ενέργεια κυρίως. Νομίζω πως όντως υπάρχει μια, ένας φραγμός στην επικοινωνία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και τους Ευρωπαίους πολίτες και είναι πιθανότατα η πιο σημαντική πτυχή για, την, για, για την, το ξεκίνημα οποιοδήποτε προγράμματος για την, για την κοινή αγορά. Ένα παράδειγμα. Όταν προτείναμε τις πρώτες 20 ανησυχίες των πολιτών, το είπαμε γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν ε, άσκοπο να πούμε εμείς ε, ποιε νομίζαμε ότι ήταν οι προτεραιότητε. Θέλαμε να ξέρουμε ποιε ήταν όντω οι προτεραιότητε. Είπαμε πρέπει να πάμε στους καταναλωτέ, να πάμε στους πολίτες και να δούμε ακριβώς ποιε είναι οι στόχοι. Και το κάναμε με πολύ συγκεκριμένο στόχοθετημένο τρόπο. Μερική απάντηση είναι ότι η Κομισιόν πρέπει συγκεκριμένα να κάνει κάτι επί τις ιδίες βάσεις όπως κάνουμε για τις 20 ε, μεγαλύτερες ανησυχίες, να πάει δηλαδή σε διάφορα κανάλια να απευθυνθεί άμεσα στους καταναλωτές, να πάρει τις απαντήσεις τους, να αναλύσει αυτές και μετά να επανέλθει και να μας πει ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρώτο. Και μετά το δεύτερο είναι ότι η Κομισιόν θα πρέπει πραγματικά να ιδιοποιηθεί την υπόθεση αυτή έτσι ώστε οι πολίτες και οι καταναλωτές να θεωρηθούν ως αναπόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε πολιτικής. Εάν αυτό το θέσουμε σε εφαρμογή σε όλες μας τις νομοθεσίες, νομίζω πως θα έχουμε πολύ προχωρήσει ώστε να λύσουμε κάποια στιγμή αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, Μονίκ. Και ένα λεπτό, ο Τζεράρτ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το φόρουμ για την ενέργεια του Λονδίνου είναι ένα καλό παράδειγμα μιας επιτυχημένης υπόθεσης, γιατί αρχικά ήταν ένα ετήσιο, μια ετήσια εκδήλωση όπου οι διοργανωτές καλούσαν τις ενώσεις των καταναλωτών γιατί είναι ευγενικό και μετά όμως κάτι συνέβη εκεί. Η DG Sanko δούλεψε πολύ σκληρά ε, και τώρα έχει φτιάξει ένα συγκεκριμένο ραντάρ και μαζί με τους ε, ε, νομοθέτες, με την DG Ενέργεια, την DG Sanko, έχουμε μόνιμο διάλογο, γιατί μία συνεδρίαση δεν δεν κάνετε διαφορά. Υπάρχει όμως συμμετοχή των καταναλωτών, συμβολή των καταναλωτών στην πολιτική ενέργεια και αυτό θα πρέπει να γίνεται σε κάθε πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έχω ακόμα 15 δευτερόλεπτα και να απαντήσω και μια ερώτηση που δεν μου ετέθη. Θα ήθελα να πω ότι το να φτάσει κανείς στους καταναλωτές <clears throat> δεν είναι εύκολο. Είναι η καθημερινή μας δουλειά ως ενώσει καταναλωτών. Πολύ δύσκολο να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για πολύ τεχνικά θέματα και μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Uh, ο Ζεράρντ Γκράφ. Ναι, η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είμαστε καλοί ε, στην... Ε, επικοινωνία. Δηλαδή, τι κάνουμε που τους ωφελεί συγκεκριμένα. Υπάρχουν μερικά λίγα παραδείγματα όπως η περιαγωγή στα κινητά, αλλά εν γέννη δεν κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Γιατί πολλά από την εσωτερική αγορά ωφελούν τον καταναλωτή. Και φυσικά αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Είμαστε πολύ μακριά από την καθημερινή ζωή των πολιτών και των πολιτών και των καταναλωτών, με συγχωρείτε. Ε, και πρέπει αυτή την ευθύνη να την μοιραστούμε όλοι. Θέλουμε να τοποθετήσουμε τον καταναλωτή, πρέπει να τοποθετήσουμε τον καταναλωτή σε πιο κέριο σημείο. Διαρκώ παίρνουμε διαμαρτυρίε γιατί δεν μπορούν να έχουν ας πούμε, μια συγκεκριμένη υπηρεσία το ίντερνετ, γιατί δεν μπορώ να κατεβάσω ας πούμε, γερμανικά ηλεκτρονικά βιβλία στην Ισπανία. Παράδειγμα, αυτά τα πολύ πρακτικά προβλήματα χρειάζεται να τα αναλύσουμε καλύτερα και να τα χειριστούμε, να τα αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό είναι πολύ καλό που φτιάξετε τα 20 πρώτα, τις 20 πρώτες ανησυχίες, αλλά πρέπει να βρούμε και τις λύσεις στα προβλήματα, που υπάρχουν λύσεις αλλά χρειάζεται να υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση και πολιτική πίεση. Ευχαριστώ, Τζέρντ. Ο κύριος Μάντερς θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Μια απλή ερώτηση. Η ερωτήση μου είναι πάντοτε απλέ. Για να απλοποιηθεί η επικοινωνία και η ροή των πληροφοριών προς τους καταναλωτές, κατά τη γνώμη μου όλοι οι καταναλωτές είναι ισότιμοι πολίτες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λοιπόν διαρκώς ε, εστιάζουμε την προσοχή μας σε οδηγίες και όχι σε κανονισμούς. Γιατί ε, αναφέρθηκε ότι ε, στους κανονισμούς το roaming περιαγωγή είναι μια από τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες που έγιναν αντιληπτέ και στου καταναλωτέ. Αλλά μένουμε στι οδηγίε όμω. Και τα κάτι μέλη καταχρώνται τι οδηγίε για να εισάγουν, να επανεισάγουν προστατευτισμό Πράγμα το οποίο ε, μπερδεύει τους κατανοητέ. Αν θέλουμε λοιπόν να του αντιμετωπίσουμε πιο ισότιμα θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή σε κανονισμού. Και γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Όπω Όπως έχω προπεί, εκεί που χρειάζεται φτιάχνουμε κανονισμούς και όσο γίνεται περισσότερο. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε στους υπερβολικούς κανονισμούς. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω όταν υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα παρεμβαίνουμε με έναν ισορροπημένο κανονισμό. Νομίζω πρέπει να ολοκληρώσουμε μια, αυτή την πολύ πλήρη συζήτηση. Εγώ αυτά που με εντυπωσίασαν ήταν η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη πολιτική. Αυτό προέκυψε από όλες τις συνεδρίες και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση για μια ρεαλιστική και ολοκληρωμένη πολιτική από την άποψη του καταναλωτή. Όλες οι ενέργειες, είτε είναι ασφάλεια, είτε είναι ανάκαμψη, είτε είναι επιβολή, είτε είναι παιδεία, ενημέρωση, θα πρέπει να είναι τμήμα μιας, μιας των ίδιων των καταναλωτών, δηλαδή των δυνατοτήτων τους, των, ε, δυνάμεών τους, των γνωστικών τους, ε, περιορισμών ή δυνατοτήτων. Εγώ στην έρευνα περί χειραφέτησης συμμετείχα και είμαι βέβαιος ότι τα επίπεδο δεξιοτήτων σε αυτή την αίθουσα τώρα είναι πολύ ψηλότερη από ότι ο μέσος όρος των καταναλωτών για τους οποίους φτιάχνουμε αυτές τις πολιτικές. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να φτιάχνονται οι πολιτικές με ένα διαφορετικό σύνολο ανθρώπων ε, υπόψη από ότι εμείς που είμαστε σε αυτή την αίθουσα. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοούμε τις δυνατότητες και πιστεύω πως έτσι θα μπορούμε να φτιάξουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική με συμμετοχή των καταναλωτών. Ευχαριστώ και σας επιστρέφω το λόγο, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Ντέιβιντ. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σου, στον, από τη νέα σου ιδιότητα, γιατί σίγουρα θα θελήσεις να ε, συμμετέχει στις εργασίες στο κοινό ερευνητικό κέντρο. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στη τελευταία συνεδρία. Τώρα έχουμε κλείσει τον κατάλογο των ομιλητών. Έχουμε ένα-δύο ομιλητέ για τη τελική συνεδρία, γιατί πρέπει να τελειώσουμε στις 12.30 ακριβώς. Και ευχαριστώ και τους διερμηνείς που μας στηρίζουν σε όλα αυτά. Και να πω ότι παρακαλώ για την τελική αυτή συνεδρία, μήπως μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο αργά για να βοηθήσουν και τους διερμηνείς. Με χαρά λοιπόν σας παρουσιάζω το τελευταία, την τελευταία προσκεκλημένη συντονίστρια για την ε, τελευταία αυτή συνεδρία. Είναι η Ναταλή Ομομπόνο, που είναι Γενική Διευθύντρια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, τα θέματα καταναλωτή και τον έλεγχο απάτη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας. Νομίζω πως η σχέση μεταξύ πολιτικής καταναλωτή και οικονομία προέκυψε σαφώς από την συνεδρία αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να θυμίσω τη σύστασή σας μιλώντας αρκά χωρίς όμως ταυτόχρονα να πάρω πολύ χρόνο. Ο τελευταίος ε, γύρος αυτός ε, έχοντας εξετάσει το θέμα της νομοθεσίας και τους μηχανισμούς προσφυγής αφορά δύο πυλώνες της ατζέντα των καταναλωτών που αναφέρθηκαν και από τον Επίτροπο Ντάλης αυτό το πρωί δηλαδή να ενδυναμωθεί η αποτελεσματικότητα του σεβασμού της πρόσβασης των καταναλωτών και να έχουν αποτελεσματικές ε, δυνατότητες προσφυγής οι καταναλωτές όπου χρειάζεται όπως ελέγχθη σήμερα το πρωί, δεν ακεί να υπάρχει ένα τέλειο κτίριο νομοθεσίας που αναφέρεται στα δικαιώματα και στις ε, υποχρεώσεις όλων, θα πρέπει όμως να τη χάνει και σεβασμού ταυτόχρονα και θα πρέπει οι καταναλωτές να μπορούν να βρουν το δικαίωτο τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό ρόλο τη Γενική Διεθνή του Ανταγωνισμού και ε, προστασίας του κατανοητή τις οποίες έχουμε και είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί είμαι πεπισμένη ότι η αποτελεσματικότητα συγγνώμη, μιας πολιτικής κατανάλωσης περνάει και από την κατανάωση και καλή εφαρμογή της νομοθεσίας και από τους νόη και από τους δε. Παραδείγματο χάνει καθ' όλη τη διάρκεια του έτος στην Εθνική Επικράρεια 2.500 περίπου ελεγκτές ελέγχουν στην Γαλλία βέβαια, αλλά αυτή η εμπιστοσύνη που δίνεται στους καταναλωτές στην στο εθνικό τους κράτος είναι σημαντική για να αποκτήσουν και εμπιστοσύνη γενικά όταν ε, εμπορεύονται εκτός συνόρων. Σήμερα έχουμε πολλές δυνατότητες για να ελέγχουμε το θέμα της εφαρμογής των νόμων. Τις εθνικές αρχές, σε κοινοτικό επίπεδο κοινέ δράσεις ε, συνεργασίας με τις εθνικές αρχές, το δίκτυο δηλαδή CPC, που έχει σαν στόχο να εξασφαλίζει στους ε, Ευρωπαίους καταναλωτές ε, όταν αγοράζει ένα αγαθό υπηρεσία εκτός των συνόρων τους το σεβασμό της νομοθεσίας υπάρχουν οι λεγόμενοι που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχουν οι αρχές ελέγχου. Επίσης, Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο των Καταναλωτών. Υπάρχει, όπως θα μας εξηγηθεί σε λίγο, υπάρχουν, λέω, διατάξεις και διαδικασίες ε, για την επίλυση των προσφυγών εκτός ε, εξωτικά, δηλαδή πολλές φορές πρόκειται για μικρά ποσά και κανένας ε, καταναλωτής δεν θέλει να ξεκινήσει με μία ε, ε, προσφυγή στη δικαιοσύνη για να επικρατήσει το δίκαιό του. Γι' αυτό υπάρχουν για τους καταναλωτές αποτελεσματικοί μηχανισμοί για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα εκτός ε, δικαστηρίου. Να ζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα του ελέγχου της αποτελεσματικότητας του νόμου, το τα μέσα που έχουν οι καταναλωτέ στα χέρια του για να πετύχουν αυτό και θα έχουμε τρεις ομιλητέ. Η κυρία Ρόζα Τούν, Ευρωπαία Βουλευτή, μέλος της Επιτροπής ΙΜΚΟ του Κοινοβουλίου, που έχει προετοιμάσει μία έκθεση για το Internal Market Scoreboard την Ιάρα του 2010 και επίσης και ένα ψήφισμα για τις διαφωνίες online. Η κυρία Ιτραπέλ μας, ε, διευθύντρια του ε, κρατικού οργανισμού καταναλωτών του Βελγίου, που θα σας παρουσιάσει τις εμπειρίες της και τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών και ο Σεβικέ από την ε, Δανική Ένωση Καταναλωτών που ασκεί το αξίωμα αυτό εδώ και πέντε χρόνια έχουν περάσει από το δικαστήρι, από το Υπουργείο Συγγνώμη Δικαιοσύνης και θα σα παρουσιάσει τις εμπειρίες για την εφαρμογή των μέσων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα μιλήσει ίσως και για προτάσεις για να δοθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο ισχύον διατακτικό. Θα ήθελα λοιπόν αμέσως να δώσω το λόγο στην κυρία Ρόζα Τουν υπενθυμίζοντας ότι σας καλώ όλους να συμφιλώσετε δύο στόχους μάλλον να συμφιλώσετε δηλαδή να μην ε, ε, ε, να μην θυσιάσουμε το χρόνο που πρόκειται να αφιερθεί στη συζήτηση, ο καθένα δηλαδή να μην μιλήσει πάνω από τρία λεπτά. Απ' την άλλη μεριά να μην μιλάτε τόσο γλυκόρα που οι διερμηνεί να μην μπορούν να σα παρακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ακούσαμε το εξή ότι οι καταναλωτές δεν θέλουν επανόρθωση μερικές φορές γιατί δεν αξίζει την ταλαιπωρία. Και συνεχίζω στα πολωνικά, λέει ο Μιλήτρια. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και χαίρομαι που κάποιος το είπε. Στην πραγματική ζωή, αλλά και στην εικονική, αυτή είναι η κατάσταση. Οι καταναλωτές δηλαδή δεν ε, κάνουν διασυνοριακές αλλαγές ισπανίως γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη και γιατί μπερδεύονται με τις διαφορετικές γλώσσες και τους διαφορετικούς κανόνες. Νιώθουν ε, δηλαδή αβοήθητοι. Όλοι έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Εμείς ως Ευρωβουλευτές συχνά ταξιδεύουμε. Αγοράζουμε εισιτήρια, ακυρώνεται μια πτήση στο αεροδρόμιο για παράδειγμα. Έχουμε όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, ταξιδιωτών ε, μια καλή ρύθμιση. Αν όμως ακυρωθεί η πτήση μας, εκεί ε, κάπως νιώθουμε αβοήθητοι. Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες αποφασίζουν και μας στέλνουν κάπως αλλιώς τον προορισμό μας ανάλογα με το πώς τις βολεύει εκείνες και όχι όπως βολεύει εμάς. Έχω δουλέψει πάνω στην επίλυση διαφορών online. Έχω δουλέψει λοιπόν πάνω στην οδηγία αυτή και μπορώ να σας πω ότι τα βήματα τα οποία αναλαμβάνονται προκειμένου οι καταναλωτές και οι εταιρείε να μπορούν πιο εύκολα να λειτουργήσουν μέσα στην εσωτερική αγορά. Αυτά λοιπόν ε, τα βήματα που έχουμε κάνει είναι μικρά βήματάκια. Πάντα με μικρά βήματα. Ε, έτσι χτίστηκε και η Ευρώπη. Αλλά θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Και θέλουμε να ενισχύσουμε και την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Για να ε, τα πετύχουμε όμως όλα αυτά, χρειαζόμαστε λύσεις οι οποίες να είναι εύχριστες εύκολα κατανοητές, με διαφάνεια και που να μην προορίζονται σε αυτούς που τα συνέταξαν, αλλά να προορίζονται για χρήση των καταναλωτών. Πρώτα απ' όλα λοιπόν αυτό που είναι για μένα σημαντικό είναι ότι τα έντυπα, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίλυση διαφορών μέσω του διαδικτύου θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητά και να έχει εύκολα πρόσβαση σε αυτά ο κόσμος. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνεται. Δηλαδή στο πόρταλ της Ευρώπης να μπορεί κανείς πατώντας ένα κουμπί να ενημερώνεται για αυτά τα πράγματα και πρέπει να υπάρχουν λίγες πηγές, λίγα link από εκεί και πέρα, γιατί δεν πρέπει να μπερδεύεται ο καταναλωτής, θα πρέπει εύκολα να μπορεί να βρίσκει αυτό που θέλει. Και πρέπει να υπάρχει και μια διευκόλυνση coaching, να μπορεί δηλαδή να ζητήσει βοήθεια. έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα να καταλάβει ο καταναλωτής τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Και να μπορούν ε, αυτές, ε, αυτή η διαδικασία επίλυση διαφορών μέσω του διαδικτύου να χρησιμοποιείται και σε εσωτερικό επίπεδο και διασυνοριακά. Ίσως να πρέπει η πλατφόρμα η ίδια στο διαδίκτυο, η οποία αναφέρεται στην ε, επίλυση αυτή διαφορών ε, μέσω διαδικτύου, να αναφέρει ποιες είναι οι δυσκολίες με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπος ο καταναλωτής. Ευχαριστούμε η κυρία Άπελμανς τώρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών. Πολλά θα είχα να σας πω, αλλά θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα τρία λεφτά που μου δώσατε. Ο καταναλωτής όταν αντιμετωπίζει θέματα επίλυσης διαφορών διασυνοριακά δεν μπορεί από μόνος του να το κάνει. Πρέπει να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών, ο οποίος θα αναλύσει την ε, κατάσταση και θα απευθυνθεί στο αντίστοιχο κέντρο καταναλωτών της χώρας από την οποία αγοράστηκε το προϊόν. Ερχόμαστε σε επαφή δηλαδή και έτσι προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Αυτά κάνουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών. Είμαστε δηλαδή η γέφυρα ανάμεσα στον καταναλωτή και τον πολιτή. Ακριβώς γιατί υπάρχουν διαφορετικές συνήθειες και διαφορετική νομοθεσία πολλές φορές στις διάφορες χώρες. Έχουμε αντιμετωπίσει 30.000 ε, ε, περιπτώσεις και έχουμε απαντήσει σε 80.000 ε, περιπτώσεις. Έχουμε μια αύξηση 24% από το 2007. Σε 40% των ε, προσφυγών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών βρέθηκε ε, φιλικά λύση. Σε 13 περιπτώσεις ε, χρειάστηκε να πάμε στις αναλλακτικέ μεθόδους επίλυσης διαφορών και στις 46% των περιπτώσεων δεν βρέθηκε λύση. Και αν ε, ο πολιτής δεν συμφωνήσει για την διευθέτηση, παρόλο που ο νόμος λέει ότι πρέπει, οφείλει, τότε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα. Τότε συμβουλεύουμε τον καταναλωτή να προσφύγει στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών. Αν για την περίπτωσή του δεν υπάρχει, τότε το συμβουλεύουμε να ξεκινήσει άλλη διαδικασία δικαστική. Βέβαια, περισσότεροι καταναλωτές δεν θέλουν να μπουν σε τέτοιες διαδικασίες. Οι συλλογικέ προσφυγές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να ξεκινήσουν μια δικαστική διαδικασία. Υποστηρίζουμε επίση την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια οδηγία όσον αφορά τι αλλακτικέ μεθόδου επίλυση διαφορών. Το κέντρο μα συνεργάζεται στενά και με το CPC και με τα Εθνικά Σώματα επιβολή του Νόμου. Μόνο με την επιβολή του νόμου μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους καταναλωτές. Αλλά τα δίκτυα καταναλωτών ζητούν έλεγχο σε εθνικό επίπεδο ε, μέσω ενό ε, σώματο που να διέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία για το ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή. Είμαστε δίπλα στον καταναλωτή, τον ενημερώνουμε για τα δικαιώματά του και τον βοηθούμε να επιλύει τι διασυνοργικές του διαφορέ. Χρειάζεται εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά και γι' αυτό φροντίζουμε και εμείς. Είναι ζωτική σημασία. Τέλος, χάρη στην ε, καταγραφή όλων των περιπτώσεων, έχουμε μια βάση δεδομένων λοιπόν, οπότε ο Ευρωπαίος νομοθέτης βρίσκει εκεί στοιχεία για να εκπονήσει καλύτερη νομοθεσία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, έχω κάποιες διαφάνειες, οπότε παρακαλώ να μου τις δείξετε. Ας αρχίσουμε από την αρχή παρακαλώ με τις διαφάνειες. Θα μιλήσω για την επιβολή και όπως είπε και η Επίτροπος Ρέντινγκ σήμερα το πρωί, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, τουλάχιστον αυτό λέει δικιά μου η εμπορία, είναι ότι δεν είναι εύκολη η ζωή για τον απλό καταναλωτή που δεν ξέρει απονομικά, ούτε βέβαια και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι νομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κανόνες. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να ενισχύσουμε την επιβολή διασυνοριακά. Θα σας πω δύο λόγια. Τι γίνεται όταν υπάρχει έλλειψη συνοχή στην νομοθεσία, που χρειαζόμαστε περισσότερη αναρμόνιση, και ποιοι κανόνες πιστεύουμε ότι είναι ξεπερασμένοι. Και το τελευταίο που θα σας πω είναι ένα πρόγραμμα εργασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τη μια μεριά, ο Ευρωπαίος καταναλωτής ε, χαίρει διαφόρων ε, δικαιωμάτων. Μπορεί να βασιστεί σε κανόνες που επιβάλλουν την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν στη χώρα του. Μπορεί να πάει και στο δικαστήριο της χώρας του. Βέβαια αυτό δεν το έχω δει ακόμα έρχονται ακόμα και νομικοί καθηγητές που έρχονται σε μένα και ζητάνε τη βοήθειά μου. Γιατί τι συμβαίνει. Δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Γιατί ε, τα άτομα δεν θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον μιας πολυεθνικής. Μπορεί να πάνε στις εφημερίδες ή μπορεί να πάνε στον ομπουτσμαν ε, για τους καταναλωτές. Οπότε τι γίνεται. Εμείς προσπαθούμε να επιβάλλεται ο νόμος στη χώρα του πολιτή η σχετική νομοθεσία βασίζεται στην προέλευση του πολιτή. Δηλαδή ο νόμος που εφαρμόζεται είναι εκείνος που ισχύει στη χώρα του πολιτή. Έχουμε όμως το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα δεν έχουμε εναρμόνιση όσον αφορά τις ε, αποζημιώσεις. Άρα δεν μπορούμε να αισθήσουμε αποζημίωση. Έχουμε επίσης ελάχιστη εναρμόνιση σε πολλούς τομείς πράγμα το οποίο οδηγεί σε διαφορά στο βαθμό προστασίας και άρα δεν είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του νόμου. Προτείνω λοιπόν δύο πράγματα για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Πρώτον, περισσότερη εναρμόνιση. Και σε ορισμένους τομείς χρειαζόμαστε και πλήρη εναρμόνιση. Τώρα έχουμε την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών που έχουν πλήρη εναρμόνιση όσον αφορά τις απαιτήσει υποχρεώσεων για την απόσυρση, αλλά το χρειαζόμαστε και για τις επανορθώσεις. Ή πρέπει να βάλουμε και μια ρήτρα η οποία υποχρεώνει τους πολιτές να λαμβάνουν υπόψη τους και το τι ισχύει στη χώρα του καταναλωτή. Πρόγραμμα εργασίας. Κοιτάξτε, θα είμαι εδώ σύντομο. Ε, τίμασα κάτι που λέει εδώ τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε και κοινού κανόνες στην δημοσίευση, γιατί δεν είναι πάντα οι ίδιοι. Και αυτό προσθέτει παραπάνω δυσκολίες στους καταναλωτές που έχουν να κάνουν επιχειρήσεις που δεν τηρούν το κανόνα. Οπότε, μια γενική ρήτρα που είναι υποχρώνει τις επιχειρήσεις, τις διάφορες συμβατικές σχέσεις, να σέβονται την νομοθεσία της χώρας του καταναλωτή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες που είναι ξεπερασμένοι. Εμείς ετοιμάζουμε καταθετήριες γραμμές για ε, τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook για παράδειγμα. Και αν δείτε την οδηγία του 2002 ο ορισμός εκεί μιλάει για την αποστολή μηνυμάτων. Ναι, αλλά τεχνικά δεν στέλνουμε μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, παίρνουμε μηνύματα. Οπότε αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή πρέπει να δούμε και τους κανόνες αυτούς που είναι ξεπερασμένοι. Πριν από λίγα χρόνια το διαδίκτυο ήταν εντελώ διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Οπότε πρέπει να γίνει και αυτό αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην επιβολή του νόμου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν, έχω μια πληροφορία που ίσως να σας απογοητεύσει, ότι δηλαδή, εάν δεν θέλουμε πολύ να καθυστερήσουμε, δεν θα έχω τη δυνατότητα να δεχτώ ερωτήσεις από το ακροτήριο. Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη σύνοψη των παρεμβάσεων που έγιναν, ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι η εσωτερική η αγορά παίρνει φυσικά χρόνο και είναι μια καθημερινή εργασία στην οποία επιδίδεται η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο με διάφορους ε, σημαντικούς βεβαίως φορείς ε, για να το στηρίζουν. Να τονίσουμε φυσικά το σχέδιο οδηγία για την ε, εναλλακτική επίλυση των διαφορών ή για την online επίλυση διαφορών. Άλλο παράδειγμα, η τακτική επανεξέταση κειμένων, νομοθετικών κειμένων και από αυτήν την άποψη ακούσαμε μια έκκληση για ενίσχυση των τρόπων δράσης των αρχών ελέγχου ε, για να επιβάλλουν το σεβασμό των ε, δικαιωμάτων του καταναλωτή μαζί με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή κτλ. Αλλά το ερώτημα που θα μπορούσε κανείς να θέσει σήμερα είναι ποιος είναι ο βαθμός γνώσης ε, που έχουν οι καταναλωτές για το σύνολο των θετικών υπηρεσιών. Ε, και αυτό είναι μια δουλειά, για την, ένα έργο προς το οποίο θα πρέπει να εμβαθύνουμε νομίζω όλοι. Πάολα, θες να προσθέσεις κάτι? Ναι, τρία δευτερόλεπτα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Μάλκομ και όλους τους συμμετέχοντες γιατί νομίζω πως η σημερινή συζήτηση έδειξε πόσο δουλειά έχουμε ακόμα να κάνουμε στον τομέα του καταναλωτών. Η Επίτροπος και Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ ε, είναι πολύ σημαίνει σε αυτό το θέμα. Έχουμε φτιάξει μια ατζέντα, ένα είδο μανιφέστου του τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε αποδείξει πόσο σοβαρή είναι η Κομισιόν για τα ενδιαφέροντα τα συμφέροντα των καταναλωτών και εν γέννη για τον καταναλωτή ως σημαντικό και θεμελιώδες τμήμα της ε, εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Ωραία. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τεστόρη την κυρία Ομομπονό, τον κύριο Μέρ και όσους ε, χρειάστηκε να φύγουν και να εγκαταλείψουν ε, την ε, αίθουσα. Πραγματικά ήταν πολύ σπουδαία η ακρόαση σημερινή. Είχαμε διακεκριμένους ομιλητές. Ελπίζω να σας ευχαριστήσω. Είχαμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σήμερα και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που μας βοήθησαν και ζητώ συγγνώμη γιατί με το ζήλο μας να πούμε όλα μιλούσαμε κάποιες φορές κάπως γρήγορα. Αλλά δεν πειράζει, μείνουν και λιμερικά για την επόμενη φορά. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλου όσου συμμετείχαν. Είμαι ευχαριστημένο που μπορέσαμε να έχουμε διάφορε παρεμβάσει από εκπροσώπου των ενώσεων καταναλωτών. Νομίζω πω ήταν καλή ευκαιρία ε, για μένα, εξ ονόματο των ε, μελών τη Επιτροπή μα, να εκφράσω την ε, επέτειο τη ενίας αγορά μου ζητήθηκε να συμβάλλω με κάποια ιδέες ώστε να φτιάξουμε ένα είδος think tank με διάφορους από εσά εκεί για το μέλλον και της, της πολιτικής καταναλωτή και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον αυτή τη ατζέντα για την καταναλωτή και είναι πολύ καλό που συμπίπτουν όλε αυτέ οι δραστηριότητε γιατί έτσι συνδυάζουμε τι ιδέε, ιδέε που προκύπτουν από αυτή την ακρόαση, στην έκθεση την Επιτροπή μα και προωθούμε αυτή τη ε, δημιουργία της ατζέντα του καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το πρόγραμμα του καταναλωτή και τα κονδύλια που θα στηρίξουν αυτή την ιδέα. Ήδη έχουμε πει πως δεν είναι πολύ συγχρονισμένο αυτό με την ε, ατζέντα του καταναλωτή, αλλά η κυρία Τεστόρη και ο κύριος Ντάλι επιβεβαίωσαν ότι αυτές οι δύο πτυχές θα είναι σωματωμένες, αλλά για δημοσιονομικούς λόγους πρέπει να προχωρήσουμε και να ε, ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα περί καταναλωτή. Μένει λοιπόν μόνο πια να ευχαριστήσω το επιτελείο της Επιτροπής, τη δικιά μας, το δικό μας επιτελείο, Τζέρετ Μπιάνκα και όπως βλέπετε συνέλεξαν τις δικές σας πληροφορίες. Συνεχίστε να στέλνετε τις ιδέες σας στην Επιτροπή μας, γιατί όπως βλέπετε η δουλειά μας συνεχίζεται. Δεν ήταν εδώ η Κομισιόν για να σας παρουσιάσει κάποια οριστικοποιημένη ατζέντα και νομίζω πως υπάρχουν πολλά σημαντικά ε, στοιχεία που θυλέξαμε σήμερα, ιδιαίτερα τα θέματα ανταγωνισμού, πολιτικής ανταγωνισμού αποκτούν ε, μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα γιατί οι online επιχειρήσεις και το εμπόριο online δημιουργούν νέε προκλήσει. Και είμαι ευτυχή που η κυρία Κρόζ συμμετείχε σε αυτή την, την, την ακρόαση, γιατί στην πρόσφατη έκθεση, μάλλον ανακοίνωσή της, μίλησε για τα σήματα, τα εμπορικά σήματα στο online εμπόριο και τη σημασία αυτών. Πάντως, σίγουρα πρέπει να βασιστούμε σε μια πλατφόρμα εμπειρίας και γνώσης και η συνεργασία μας νομίζω συμβάλλει στη δημιουργία αυτού. Και ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν. Νομίζω πως θα πρέπει με ένα θερμό χειροκρότημα να ευχαριστήσουμε όλους τους ομιλητές. Σας εύχομαι καλό, καλή όρεξη και καλό απόγευμα. Και ευχαριστώ και όσους ήταν online και συμμετείχαν ε, από μακριά στη συνεδρίασή μας.